καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση για την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Κωνστάνσιο, να ξεκινήσουμε με τη μερίσια διάταξη. Εγκρίνεται ε, η μερίσια διάταξη. Υπάρχουν σχόλια, διαφωνίες, όχι. Πάμε σε ανακοινώσει του Προέδρου, το τι γίνεται με τις οργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Το πρώτο αφορά το θέμα της ε, τιτλοποίησης. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε στις 28 Μαρτίου και σημειώθηκε πρόοδος για τα STS ε, και του CRR. Στο θέμα του STS το αποτέλεσμα ήταν το εξής. Οι συνομοθέτες συζήτησαν το έγγραφο της Κομισιόν για τα επιλέξιμα μέρη στην ε, αγορά τίτλοποίησης και τα κριτήρια ομογενοποίησης σύμφωνα, σύμφωνησαν να δώσουν έντολη στην Κομισιόν να συνεχίσει την ε, πρότασή της και να προτείνει μια διατύπωση για τα κριτήρια ομογένειας, ομοιογένειας με βάση τα όσα ακούστηκαν στην συνεδρίαση. Επίσης προτείνουμε να υπάρξει ένα σχέδιο stress test με βάση τα όσα ισχύουν από την νομοθεσία. Πέρα από τις απαιτήσει, πέρα από αυτά, συμφωνήθηκαν κάποιες απαιτήσει για την δέουσα επιμέλεια. Και τέλος, ε, τέθη το ζήτημα της απαγόρευσης έπανα και τίτλοποίησης. Το θέμα του ΣΥΑΡΑ, το αποτέλεσμα ήταν το εξή για την ε, εντολή της ε, EBA για να μπορέσει να καθορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις με βάση την εσωτερική αξιολόγηση. Υπήρξε μια συμφωνία, όπως επίσης και για την χρήση δεδομένων όπου αυτό απαιτείται. Επίσης εξετάστηκε περαιτέρω το ζήτημα της ε, τίτλοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπό συγκεκριμένε συνθήκες θεσμικές εγγυήσει για την εγγύηση τέτοιων συναλλαγών. Ζητήθηκε από την Κομισιόν να αξιολογηθεί κατά πόσον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μέτρα τα οποία εξομοιώνονται προς ε, μερίσματα μετρητών. Τέλος, συμφωνήσαμε σε κάποια άλλα πολιτικά ζητήματα για να ευθυγραμμιστούμε όσο δυνατόν περισσότερο με το σχέδιο της Επιτροπής της Βασιλείας και οι συνομοθέτες ενέκαναν κομμάτι των τεχνικών εργασιών. Αυτά για τον πρώτο τριμερή διάλογο και έχουμε και τον δεύτερο που αφορά την πέμπτη αναθεώρηση της οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος που έλαβε χώρα στις 4 Απριλίου και είχαμε έξι ζητήματα. Τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Θα επανέλθουμε σε αυτές τις προσεγγίσεις ενώ η Κομισιόν θα αναφέρει για τους πιθανούς δρόμους που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Δεύτερο ζήτημα, η μονάδα οικονομικών πληροφοριών και η Κομισιόν και το Συμβούλιο συμφώνησαν στην ανάγκη αυξημένη συνεργασίας. Ε, η Κομισιόν συμφώνησε να δώσει κάποια σχέδια διατύπωσης. Ε, το θέμα των αξιοπινών πράξεων. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα των ορίων για τις αξιοπινές πράξεις. Για τις προπληρωμένες ε, κάρτες ανατέθηκε στην ομάδα εργασίας να βρεθεί μια λύση. Πέμπτο, κυρώσεις. Είπαμε πως το Συμβούλιο ήταν ανοιχτό σε κάποιες προτάσεις του Κοινοβουλίου. Και τέλος, εντολή για τεχνικές εργασίες ε, που έγιναν την επόμενη μέρα στις 5 Απριλίου σε όλα τα ζητήματα που αναφέραμε. Ο τριμερής διάλογος θα συνεχιστεί τον επόμενο μήνα στις 10 Μαΐου. Αυτά για τον τεχνικό τριμερή διάλογο. Και τώρα μπορούμε να πάμε στο βασικό θέμα της ημέρας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε και βεβαίως ε, μενουμε την συνήθη συζήτησή μας και την ετήσια έκθεση, την ετήσια η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγα λεπτά στο site της ΕΚΤ καλύπτει τις οικονομικές πολιτικές εξελίξεις το 2016 και τις τρέχουσες δραστηριότητες του ευρωσυστήματος στους διάφορους τομείς αρμοδιότητας του επιπλέον. Έχουμε βεβαίως και στις 4 Απριλίου την ε, έκθεση την οποία έστειλε ο πρόεδρος Δράγκη στον πρόεδρο Ταγιάννη και έχουμε βεβαίως και τα σχόλια στην έκθεση του 2015. συγητής ήταν ο Ραμόν Τρεμόζα. Αυτά σας τα έστειλε η γραμματεία το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και σύμφωνα με το άρθρο 284 της συνθήκης η έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κομισιόν και Συμβούλιο και η ΕΚΟΝ θα παρουσιάσει την αρχή έκθεση. Ο εισηγητής Δεν έχει καθοριστεί, θα οριστεί από τους σοσιαλδημοκράτες, αν κατάλαβα καλά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια εισαγωγική δήλωση της ΕΚΤ από τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Κωνστάνσιο. 15 λεπτά το πολύ και μετά θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. 2 λεπτά η κάθε ερώτηση, 3 λεπτά οι απαντήσεις, 5 λεπτά συνολικά. Έχουμε λοιπόν έναν κατάλογο μιλητών που έχουν ορίσει οι πολιτικές ομάδες και αν υπάρχει χρόνος θα συνεχίσουμε με τους παρόντες. Τέλειωσα εγώ λοιπόν να δώσω τον λόγο στον κύριο Αντιπρόεδρο και χαίρομαι που είμαστε πιο αισιόδοξοι τώρα γιατί πηγαίνει σχετικά καλά η ευρωπαϊκή οικονομία και θέλουμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σα για να σα παρουσιάσω την ετήσια έκθεση τη ΕΚΤ για το 2016. Η ετήσια έκθεση αποτελεί ουσιώδε στοιχείο τη δημοκρατική μα λογοδοσία. Στηρίζει τη δημοκρατική συζήτηση ω προ τη λήψη αποφάσεών μα. Και η λογοδοσία μα δεν σταματά φυσικά με την υποχρέωση υποβολή εκθέσεων. Αυτή η ευκαιρία μα εξασφαλίζει συζήτηση τη ετήσια έκθεση με εκπροσώπου των λαών τη Ευρώπη. Μάλιστα, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την λογοδοσία μα προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για την απαρχή μια ε, καλό εφαρμοσμένη ε, διαδικασίας και η σημερινή ε, ανταλλαγή απόψεων θα τροφοδοτήσει και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεση τη ΕΚΤ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μα γιατί θέλουμε να μεριμνήσουμε ότι πραγματικά ανταποκρινόμαστε στη δημοκρατική εντολή που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι ανεξάρτητη προκειμένου εντό εντολή τη να δρά χωρί πολιτικέ παρεμβολέ. Και επίση είναι δημοκρατικά και νομικά υπόλογη για να εξασφαλίσει ότι πραγματικά δρά με βάση την εντολή τη. Ω ήθιστε, σήμερα δημοσιεύσαμε και το feedback μα, το σχολιασμό μα, ό,τι αφορά το ψήφισμά σα για την προηγούμενη ετήσια έκθεσή μας θα κάνω μερικά ε, μια παρουσίαση των βασικών μας πολιτικών και το, ε, τη συμβολή του στην υλοποίηση του στόχου μα, τη διατήρηση τη της αθερότητας τιμών. Επίση, θα τονίσω τη σημασία ενό ισχυρού χρηματοπιστωτικού συστήματο ε, για την ευημερία τη Ευρωζώνης. Η ανάκαμψη τη Ευρωζώνης και η στήριξη τη νομισματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2016 ανταποκρίθηκε σε με μια πολύ απαιτητική και δύσκολη χρονιά. Την τελευταία φορά που μίλησε εδώ τον Απρίλιο πέρυσι, η παγκόσμια οικονομία ανάρωνε μετά από ένα οξύ κρούσμα χρηματοπιστωτικής αστάθειας. Αυτό το επεισόδιο μάλιστα έδωσε πάλι λαβή για μια νέα έξαρση βαθύτατη της απεισιοδοξίας, όχι μόνο για την ικανότητα της παγκόσμιας οικονομίας να περάσει σε θετική ανάπτυξη, αλλά και για την ικανότητα των κεντρικών τραπεζών να κατευθύνουν τις οικονομίες τους εφαρμόζοντας μη συμβατικά μέσα νομισματικής πολιτικής. Μάλιστα είχαμε ρεκόρ ε, χαμηλής, ε, χαμηλού πληθωρισμού με ε, απότομη πτώση των τιμών των βασικών προϊόντων. Έχει περάσει ένας χρόνος και χάρη στα μέτρα που λάβαμε τότε και μάλιστα διαψεύδοντας κάποιους σκεπτικιστές της πολιτικής μας, διαπιστώνουμε βελτίωση των μακροοικονομικών συνθήκων και πολλές χαρμόσυνες ειδήσει. Έχουν αποσοβηθεί οι φόβοι του αποπληθωρισμού και παλά μια σχετικά χαμηλή ανάπτυξη έχουμε σταθερή αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7 πέρυσι και το πρώτο τρίμηνο του 2017 η οικονομική αίσθηση έχει ανέβει στα υψηλότερα ποσοστά αυτά του 2011. Μάλιστα η ενεργεία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της από το Μάιο του 2009. Περίπου 4,5 εκατομμύρια περισσότεροι συμπολίτε μα έχουν βρει μια θέση εργασία σε σχέση με πριν από μια τριετία. Τα μέτρα μα επίση μείωσαν τον κατακαιρματισμό μεταξύ των κρατών μελών. Και η διαφορά μεταξύ ε, ε, του, της αύξησης του ΑΕΠ και των ποσοστών πληθωρισμού είναι χαμηλότερη σε σχέση με την αρχή της νομισματικής ένωσης. Οπότε τα μέτρα του περασμένου Μαρτίου δημιούργησαν πραγματικά ενάψματα νομισματικά και οικονομικά και δημιούργησαν ένα πραγματικά σημαντικό προφυλακτήρα για την ανάκαμψη της οικονομίας προκειμένου να γίνει πιο ανθεκτική σε εξωτερικές κραδασμούς και αβεβαιότητε. Το Δεκέμβριο του 2016 αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την αγορά περιουσιακών στοιχείων μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 με μειωμένο ρυθμό 60 δις ε, το μήνα από τον Απρίλιο του 2017 και μετά. Ε, ε, με, σε ευθυγράμμιση με τους μειωμένους κινδύνους σταθερότητα των τιμών. Έτσι εξασφαλίζει τις οικονομικές συνθήκες που είναι επίσης απαραίτητε ε, για να ενισχύσουν την επαναφορά του πληθωρισμού σε επίπεδα γύρω στο 2% μέσω πρόθεσμα. Τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το Μάρτιο του, το Μάρτιο του 2016 στήριξαν και τη βελτίωση των οικονομικών συνθήκων. Έχουν διευκολύνει την σταθερή μείωση της, ε, των, ε, των σύνθετων ε, ποσοστών δανεισμού των τραπεζών και των ποσοστών για δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες και ενικόθηκα δάνεια που έχουν μειωθεί σε επίπεδα ιστορικά και από το Μάιο του 2014, δηλαδή αμέσως πριν την υποβολή των αποφάσεων μας για, το, για, την ε, επιπλέον μέτρα νομισματικής πολιτικής προκειμένου να στηρίξουμε το δανεισμό στην, στην πραγματική οικονομία, η μείωση των επιτοκίων σε τραπεζικό δανεισμό έχουν φτάσει μέχρι στο 120 βασικά, βασικές μονάδες για δάνεια προς τις επιχειρήσεις, 110 βασικές μονάδες σε δάνεια προς τα νοικοκυριά και μάλιστα οι όγκοι δανεισμού έχουν ε, αυξηθεί σημαντικά ε, καθώς έχουμε αύξηση των δανείων στις εταιρείες 2% το Φεβρουάριο του 2017 από το μείον 2,9% το Μάιο του 2014 και για τα νοικοκυριά αύξηση 2,3% από μείον 0,1% ε, που είχαμε για την ίδια περίοδο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρωζώνης, έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερως από τις αλλαγές αυτές. Η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση έχει βελτιωθεί αισθητά και το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί περίπου κατά 40 βασικές μονάδες από το Μάρτιο του 2016 και γύρω στις 180 βασικές ε, μονάδες από το Μάιο του 2014 μετα... Ε, προς τα τέλη του 2016 εδραιώθηκε η ανάκαμψη και επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς και χώρες. Μάλιστα όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή σημειώνουν ανάπτυξη. Και μάλιστα οι δείκτες του πρώτου τριμήνου του 2017 δείχνουν ότι ο ρυθμός της ανάπτυξης αυξάνεται. Βέβαια, η παρακαταθήκη της, της οικονομικής κρίσης εξακολουθεί να προσδιορίζει τις σημερινές μας επιδόσεις από πολλές απόψεις. Ε, δεδομένου του μεγάλου ποσοστού των μη αξιοπιθέντων προών, ο βασικός πληθωρισμός ε, είναι σε καθοδική πορεία και μάλιστα ο συνολικός πληθωρισμός του Μαρτίου έχει μειωθεί, από ένα, έχει μειωθεί στο 1,5 από 2% το Φεβρουάριο, ενώ ο υφέρπον πληθωρισμός έχει μειωθεί από 0,9 σε 0,7%. Είχαμε μάλιστα προειδοποίηση ότι ο συνολικός πληθωρισμός ίσως μειωθεί μετά τον Απρίλιο-Μάρτιο ως αποτέλεσμα της μειωμένης του μειωμένου στατιστικού βασικού αποτελέσματος σε σχέση με τη σύγκριση των αντίστοιχων ε, τιμών και φέτος, ειδικά λόγω των τιμών του πετρελαίου. Αλλά η μείωση της, του υφέρποντος πληθωρισμού ήταν απογοητευτικό και μάλιστα οι δείκτες ε, δεν ανταποκρίνονται ακόμη στην ανάκαμψη και μειώνουν το χάσμα της παραγωγής. Σε βάση, με βάση τις προβολές που κάναμε, προβλέπουμε το 2019 πληθωρισμό γύρω στο 1,7%. Υπό τον όρο όμως ότι ο υφέρπων πληθωρισμός θα είναι 1,8% και η αύξηση των μισθών στο 2,4%. Η προβλεπόμενη αύξηση των μισθών στο βασικό σενάριο είναι απαραίτητη για τις προβολές που έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό προκειμένου να υλοποιηθούν όλες αυτές το 2019. Επιπλέον, ενώ ο βραχυπρόθεσμος ε, προβλεπόμενος πληθωρισμός ε, είχε αύξηση λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας των τιμών, ο μεσοπρόθεσμος, η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη δεν έχει επηρεαστεί. Επίσης, η αναδική πορεία του συνολικού πληθωρισμού τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί τα μάλα από τη στήριξη της νομισματικής πολιτικής. Ενώ, λοιπόν, η νομισματική μας πολιτική είναι προσανατολισμένη κυρίως στη διατηρήση της σταθερότητα των τιμών, Έχουμε βεβαίω ω καθήκον και την ταυτοποίηση και αξιολόγηση των πιθανού αντικτύπου των συστημικών κινδύνων στη σταθερότητα τη Ευρωζώνη. Η ετήσια έκθεσή μα λοιπόν αναφέρει τέσσερι κυρίου κινδύνου. Πρώτον, η πιθανότητα μια αύξηση στα παγκόσμια ασφάλιστρα κινδύνου η οποία έχει αυξηθεί σε ένα περιβάλλον πολιτική αβεβαιότητας ε, και αυλαβου τιμολόγηση των αγορών δεύτερων μια πιθανή αρνητική ανάδραση μεταξύ χαμηλή κερδοφορια των τραπεζών εν ώψη των διαρθρωτικών προκλήσεων σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και χαμηλή ονομαστικής ανάπτυξη τρίτων, πολιτική αβεβαιότητα η οποία υποβαθμίζει τι προσπάθειε για μεταρρυθμίσει, με τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους να επανεμφανίζονται για τον δημόσιο και μη χρηματοπιστωτικό τομέα σε κάποιες χώρες. Τέταρτον, ο κίνδυνος ρευστότητας αυξάνεται πάρα πολύ, στο, ο οποίος αυξάνεται, με συγχωρείτε, στον τομέα των επενδυτικών ταμείων. Πέρα από τα συστημικά πέρα από του συστημικού κινδύνου στον συνολικό τομέα τη Ευρωζώνη, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση που προκύπτει ανά χώρα και ανά κλάδο. Στοχευμένα μακροπροληπτικά μέτρα είναι τα κατάλληλα μέσα πολιτική για να δούμε την κάθε χώρα και τον κάθε κλάδο. Όπω ξέρετε, η ευθύνη για τι αποφάσει για τα μακροπροληπτικά μέτρα τη Ευρωζώνη είναι κοινή μεταξύ εθνικών αρχών και ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε τα μακροπροληπτικά μέτρα των εθνικών αρχών για τα μέσα εκείνα τα οποία προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενίσχυσε τον ρόλο της στη μακροπροληπτική πολιτική το 2016 και επίσης ανέλαβε δράση για να βελτιώσει τη διαφάνεια. Πέραν από τις δράσεις σε κάποιες χώρες στον τομέα των ακινήτων παρατηρήσαμε ότι παραμένουν κυκλικοί συστημικοί κίνδυνοι περιορισμένοι στην Ευρωζώνη και άρα μια αύξηση σε αντικυκλικά αποθέματα κεφαλαίου στην Ευρωζώνη δεν ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν αυτό. Βεβαίως συμφωνεί και με τις αποφάσεις των εθνικών αρχών με τις οποίες έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Η διαφάνεια στον τομέα της μακροπροληπτικής πολιτικής ενισχύθηκε και με το νέο διετές μακροπροληπτικό δελτίο της ε, τράπεζας τον Μάρτιο του 2016. Η ετήσια έκθεσή μας, επίσης, εστιάζει στις δράσεις που απαιτούνται για να ξεπεράσουμε την κληρονομιά της κρίσης στον τραπεζικό τομέα. Απαιτείται αποφασιστική δράση σε κλαδικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα, οι τράπεζες πρέπει να συνεχίσουν την προσαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου τους για να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Όπως δείχνουμε σε μια ξεχωριστή ανάλυση, η οποία περιέχεται στην έκθεση, η βέλτιστη στρατηγική εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάθε τράπεζας. Και βεβαίως οι ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν και διασυνοριακές ε, συγχωνεύσεις. Δεύτερον, απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να λυθεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο βαθμός και η μακροπροληπτική φύση του προβλήματος απαιτούν μια συνολική και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως οι απαντήσεις πρέπει να ληφθούν ε, από τους ενδιαφερόμενους στο εθνικό επίπεδο, αλλά πρέπει να είναι εναρμονισμένες με βάση ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μέσω παραδείγματος χάρη εταιριών χαρτοφυλακίου για να μειωθεί ακριβώς το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ζήτημα επίσης είναι ένα ζήτημα μακροπροληπτικής ε, σκοπιάς. Τώρα, για να δούμε το ζήτημα της χρηματοπιστωτικής ρυθμίσης. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρυθμίζει το σχετικό πλαίσιο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντα υπόψη και τις μακρο και τις μικροπροληπτικές ανάγκες. Το 2016 η Επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε σε διάφορες μεταρρυθμίσεις μεταξύ των οποίων η αντιμετώπιση του κινδύνου των επιτοκίων, η επανεξέταση του πλαισίου τιτλοποίησης και βεβαίως μια προδιαγραφή για το πώς θα αντιμετωπίζεται η λεγόμενη τίλεκ, e η συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Επίσης, ε, ξεκίνησε δημόσιες διαβουλεύσεις για το πώς θα αντιμετωπίζονται οι απαιτήσει δημοσιοποίησης ε, του τρίτου πυλώνα και όσον αφορά βεβαίως το πακέτο της Βασιλείας 3, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε να υπάρξει ένα πρόγραμμα για να μειωθεί ο υπερβολικός κίνδυνος στα στοιχεία και ενεργητικού, τα οποία είναι σταθμισμένα με βάση τον κίνδυνο τον Ιανουάριο του 2017 το Διοικητικό Συμβουλίο καλωσόρισε την πρόοδο της ε, Επιτροπής της ε, Βασιλείας και βεβαίω απαιτείται περισσότερος χρόνος για να οριστικοποιήσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις αλλά αναμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο στο προσεχές μέλλον. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί το μεταρρυθμιστικό πακέτο και να μην οπισθοχωρήσουμε στην πρόοδο που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο αυτό στο διεθνές επίπεδο για να επιτύχουμε ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργεί ίσως όρους ανταγωνισμού. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια επίσης έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο με την σύσταση της Τραπεζικής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα επιπλέον μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βοηθήσει και θα συνεχίσει να βοηθήσει τις ε, δύο αυτές διαδικασίες της μείωσης ε, και τη κοινή ανάληψη του κινδύνου στο πλαίσιο τη εντολή τη ω κεντρική τράπεζα και υποπτική αρχή Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιταχυνθεί η δουλειά για ένα ευρωπαϊκό κοινό σύστημα εγγύησης ε, καταθέσεων και ένα ευρωπαϊκό κοινό ταμείο διάσωση ε, παράλληλα. Η δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής πηγαίνει προ την σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τα, μέσα, τα μέτρα μείωση του κινδύνου και αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση της ε, ρύθμισης εποπτείας ε, και διάσωσης των τραπεζών, ακόμα και αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τα επιτεύγματα αυτά στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τράπεζες θα συνοδευτούν από ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για τις χρηματοχωρές και τις ε, δημοσιονομικές υποδομές, με στόχο να υπάρξει μια πλήρης Ένωση Κεφάλαια Αγορών, μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κεντρική Τράπεζα. Έτσι θεωρούμε ότι μπορεί να αυξηθεί ο διαμερισμός ε, του κινδύνου μέσω διασυνοριακών επενδύσεων, να συνεισφέρουμε στην μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τελικά να διευκολύνουμε τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η νομική βάση για μακροπροληπτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κινδύνους προς την ε, δημοσιονομική σταθερότητα καθώς επίσης να δούμε και την μακροπροληπτική προοπτική στην ρύθμιση των μη τραπεζικών ιδρυμάτων. Τέλος, η οικονομία της Ευρωζώνης απέδειξε σημαντική αντοχή το 2016. Η ανάκαμψη προχωρά και πλέον αποκτά ορμή. Η νομισματική μας πολιτική είναι η κατάλληλη και δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή μια επανεξέτασή της όμως. Θα συνεχίσουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε σε τυχόν κράδασμους. Ενώ έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, εξακολουθούμε να δούμε εξακολουθεί να πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα την κληρονομιά της κρίσης και να ενισχύσουμε τα διαρθρωτικά θεμέλια της Ένωσης. Αύριο θα ήταν τα 97 γενέθλια του Εμιλίου Κολόμου, πρώην Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω τα όσα είπε πριν από 40 χρόνια, που έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα, όταν ένα κράτος μέλος μας ειδοποίησε για το ότι θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε πει λοιπόν ο κ. Κολομπού, δεν μπορούμε να χαλαρώνουμε όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση της Ευρώπης παρόλες τις προσπάθειές μας. Ως Ευρωπαίοι μπορούμε να έχουμε αντίκτυπο όταν καταφέρουμε να βρούμε λύσεις από κοινού στα προβλήματα των καιρών μας. Αυτές οι λέξεις μας θυμίζουν την σημασία της ευθύνης μας ως Ένωσης για να συνεχίζουμε να προσπαθούμε να επιτύχουμε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, για αυτή την ομιλία σας και για την πολύ σημαντική ιστορική παράθεση που αναφέρετε στο τέλος. Τώρα θα περάσουμε στις ερωταπαντήσεις, αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, να έχετε κατά νου ότι υπάρχει και περιορισμός χρόνου. Εκ μέρους του ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μας παρουσιάσατε την ετήσια έκθεση. Βεβαίως, ε, οι νομισματικές πράξεις της ΕΚ, τα αναμφίβολα, είχαν θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας, ε, όπως διαπιστώνουμε, ο πληθωρισμός ε, προβλέπεται να φτάσει στο στόχο της ΕΚΤ και ως εκ τούτου θα παραμείνει διαχειρίσιμος μεσοπρόθεσμα όλα αυτά βέβαια ο πρόεδρος κύριος Ντράγκη ότι είπε πρόσφατα ότι η ΕΚΤ δεν προτίθεται να αλλάξει τη δέσμευσή της, ε, τη συγκράτηση των μισθών τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2018 που θα τελειώσει η ποσοτική χαλάρωση. Παρότι η ΕΚΤ ε, γνωρίζει πολύ καλά τις επιπτώσεις που μπορούν να υπάρξουν από τα αρνητικά επιτόκια. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Πότε ακριβώ προβλέπετε ότι η Ευρωζώνη ε, θα είναι αυτοδύναμη χωρίς να χρειάζεται την υποστήριξη που έλαβε πρόσφατα και τι είδου ενέργειες μπορούμε να περιμένουμε από την ΕΚΤ, τι είδου ε, επιπτώσεις προβλέπετε εσείς ότι θα υπάρξουν ε, από την αγορά. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι Όσον αφορά την ΕΚΤ, αναφέρεται ότι ορισμένα κρατημέλη καταφεύγουν στην αγορά κεφαλαίων για να αποφύγουν τα δημόσια χρέη και διάφορα άλλα αρνητικά μέτρα και για να δώσουν όθηση στις μεταρρυθμίσεις. Και ήθελα να ρωτήσω ε, η αξιολόγηση του προγράμματος αγοράς κεφαλαίων, ε, ποιες είναι οι αρνητικές ρηπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί. Ο κ. Ντομπρόφσκης μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα ε, για τον ισοσκελισμό του προπολογισμού στην Ευρωζώνη Υπάρχουν ε, κράτη-μέλη ε, που πιστεύουν ότι αυτή είναι μια αλλαγή ε, και πάρα πολλοί μιλάνε για μια εξίσωση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και ερωτώ μήπως μπορείτε λιγάκι να μας παρουσιάσετε τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στην ΕΚΤ και τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από ένα από τις ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Ε, τώρα πώς να απαντήσω τρία λεπτά. Τέλος πάντων, θα κάνω ό,τι μπορώ. Καταρχήν, όσον αφορά στην ε, πολιτική μας ε, κατά πόσο είναι κατάλληλη όχι. Θέλω να πω εξορισμού. Εφόσον δεν έχουμε αλλάξει αποφάσεις, δεν το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι η πολιτική μας είναι σωστή. Και βεβαίως διαπιστώνουμε και εξετάζουμε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεύτερον, οι προβλέψεις που έχουμε δημοσιεύσει με τα στοιχεία που καταλήγουν σε πληθωρισμό 1,7 το 2019 Αυτές οι προβλέψεις βασίζονται προφανώς σε κάποιες παραδοχές. Και μία από τις παραδοχές είναι ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει λίγο πολύ το Γιατί σε τεχνικό επίπεδο αυτό που χρειαζόμαστε για να γίνουν αυτές οι προβλέψεις είναι σταθερή ε, ισοτιμία και παίρνουμε από τις αγορές ε, το ποιε είναι προσδοκίες για τις μελλοντικές ισοτιμίες έχουμε ε, μια καμπύλη, την ΕΟΕΣ, για το ποιες είναι οι προσδοκίες για τις ε, ε, για την εξέλιξη του overnight rate, το οποίο πειράζει πάρα πολύ τις αποφάσεις μας. Με βάση λοιπόν αυτές τις προβλέψεις, το 2020 θα είναι θετικό το αποτέλεσμα. Άρα δηλαδή υπάρχουν αυτές οι παραδοχές που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις προβλέψεις μας. Και είναι σημαντικό να υπογραμμίσει κανείς ότι αυτές οι προβλέψεις βασίζονται στο να διατηρείται η νομισματική υποστήριξη που είναι σημαντική. Όπως σας είπα έχουμε μια σχετική μείωση στην ε, στον υπέρποντα πληθωρισμό και νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση που αντιμετώπισαν και οι ΗΠΑ στην πολιτική του για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το ποσοστό ανεργία μειωνόταν στι ε, ΗΠΑ, αλλά δεν αυξάνονται οι μισθοί. Περίμεναν λοιπόν και μόλι πρόσφατα ε, προσαρμόστηκαν, ε, προσάρμοσαν του μισθού στην ανάπτυξη τη οικονομία. Και εμεί θα κάνουμε περίπου το ίδιο. Πάντω υπάρχουν αυτέ οι σχετικέ προβλέψει σχετικά με το με το κόστος μισθού, μονάδα κόστους. Με πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς κατά κύριο λόγο αγοράζουμε κρατικά ομόλογα. Αυτό ισχύει και για όλα τα άλλα εργαλεία. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, ε, καμία στρεβλή εξέλιξη. Έχουμε ένα πρόγραμμα, μικρό πρόγραμμα αγοράς εταιρικών κεφαλαίων, αλλά και πάλι σας λέω δεν υπάρχουν ε, ειδικοί κλαδικοί αγοραστές. Όσον αφορά τώρα τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και τον ενδεχόμενο εξέλιξης ε, του ESM, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Απλά ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι δυνατότητες για την Ευρωζώνη είναι αυτό που αναφέρεται σε μία έκθεση ε, των πέντε Προέδρων που και εμείς στηρίζουμε. Αυτό έχει δημοσιευτεί και εκεί δεν γίνεται λόγος για μετεξέλιξη του ESM. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η Δεσποινής Περβάνος Πέρας. Ευχαριστώ για το Δεσποινής, λέει η κυρία Πέρας. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Διαπιστώνω ε, πολλά θετικά σημεία στην ετήσια έκθεσή σας. Καταρχήν, ε, είναι μια επεκτατική συνολική αθρηστική θέση. Μειώνονται τα ελλείμματα, ε, είστε υπέρ στοχευμένων κρατικών επενδύσεων και σημειώνεται τα θετικά αποτελέσματα της ε, ευνοϊκής νομισματικής πολιτικής που ακολούθησε η έκθεση ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε και το μέλλον. Ποιο θα είναι η μελλοντική δομή της ε, χρηματοοικονομικής εποπτείας και πώς θα αναθεωρηθεί το πλαίσιο της μακροπροληπτικής πολιτικής. Θα μπορούσατε να μας ε, παρουσιάσετε τις δικές σας απόψεις για τη συζήτηση αυτή, γιατί προς το παρόν είναι ανοιχτή η συζήτηση. Έχει υποβάλει το κείμενό της για τις διαβουλεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε με ανυπομονησία και τη δική σας άποψη. Και μια συμπληρωματική ερώτηση. Ε, όπως ξέρετε, η Διεθνής Διαφάνεια δημοσίευσε μία έκθεση στην οποία αναφέρει το τον κίνδυνο σύγκρουση συμφερόντων ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρίως ε, επειδή κάποιες, α, κάποιοι κανόνες ως προς α, ε, την περίοδο που θα πρέπει να μεσολαβεί από την πάυση των καθηκόντων ενός τελέχους και την ανάληψη νέων καθηκόντων στον ιδιωτικό κλάδο, ίσως δεν συνάδει με την διοντολογία σε ό,τι αφορά τις αρχές ε, που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μπορείτε να απαντήσετε και να σχολιάσετε αυτή την ε, έκθεση της διεθνούς διαφάνειας. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις Καταρχήν ως προς την πρώτη ερώτηση, ε, δημοσιεύσαμε μια ανακοίνωση εμπεριστατωμένη και μακροσκέλη επί της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία αυτής της ανακοίνωσής μας. Καταρχήν θα θέλαμε να έχουμε μια αναγνώριση αυτού του στο, μακροπροληπτικό πλαίσιο της ύπαρξης του, του SSM, του εποπτικού μηχανισμού. Κάτι που δεν είναι σαφές, γιατί με τη δημιουργία του SSM η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αναλάβει και μακροπροληπτικές αρμοδιότητες. Κάτι που δεν αναφέρεται στο νέο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαβουλεύσεις και θα ήταν χρήσιμο για να δοθεί και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το καθεστώς μιας μακροπροληπτικής αρχής όπως ισχύει με άλλες κεντρικές τράπεζες σε χώρες μέλη όπου οι κεντρικές τους τράπεζες έχουν οριστεί ως οι αρχές ε, οι αρμόδιες για τη μακροπροληπτική εποπτεία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, επέκταση των ε, μέσων που αναφέρονται, των μέσων δηλαδή της μακροπροληπτικής πολιτικής, που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, Αναφέρουμε επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί απόλυτα ότι στο πλαίσιο της εποπτείας θα πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στα προβλήματα και τους κινδύνους αντικατάστασης και όχι μόνο μακροπροληπτικής αποπτίας. Και αυτό θα πρέπει να, ε, να επιτευχθεί με ένα σαφή επιμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της μικρο- και της μακροπροληπτικής εποπτείας. Και αυτή η διάκριση είναι σημαντική. Έχουμε πάντως δημοσιεύσει τη σχετική ανακοίνωση που είναι πολύ πιο διεξοδική και για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπω εκεί. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, ξέχασα τη δεύτερη ερώτηση. Πολύ σύντομα. Γιατί είχαμε επαφές με την διεθνή διαφάνεια με πολλές ε, συνεδριάσεις. Εμείς ε, σχολιάσαμε τις συγκεκριμένες παραγράφους ε, της έκθεσης και μάλιστα συμμετείχαμε και σε μια δημόσια συζήτηση της έκθεσης αυτής στέλνοντας ένα μέλος του, διοικητικού, του εκτελεστικού μας συμβουλίου. Και είπαμε ότι μας ενδιαφέρει ο διάλογος και είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Άλλωστε, η έκθεση της διεθνούς διαφάνειας ε, εγκομπιάζει κάποια πρόσφατα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να εγγυηθεί αυτή τη διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση, σύγκρουση συμφερόντων, θα ήθελα να πω δύο τινά. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν στις ε, συμβάσεις τους εν, μια περίοδο ενό έτου κατά το οποίο δεν μπορούν να λάβουν καθήκοντα ή ε, θέσει στον ίδιο τομέα. Τώρα, για τα υπόλοιπα ε, μέλη του Συμβουλίου Διοικητών τη Κεντρική Τράπεζα, ε, ισχύει ένα ένας κώδικα που επίση αναφέρει μία περίοδο από την οποία θα πρέπει να απόσχουν από την ανάληψη εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε χρηματοπιστωτικό κλάδο. Επίσης για το Εποπτικό Συμβούλιο η περίοδος αυτή είναι διετής. θα προβούμε σε μια διεξοδική ανάλυση όλων των στοιχείων, αλλά ισχύουν μέτρα για τα ανώτατα, τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη διοικητικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κύριος Μπένιτ και τώρα από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Κωνστανσιο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στις απαντήσεις που δώσατε στον ε, κύριο Μουρεσάν για τις προβλέψεις του πληθωρισμού. Εάν κατάλαβα καλά, οι προβλέψεις που δημοσιεύσατε βασίζονται στο ότι η μακρο, η βραχυπρόθεσμοι, τα μακροπρόθεσμα με συγχωρείτε, τα ε, επιτοκία, τα overnight rates θα παραμείνουν σταθερά. Οπωσδήποτε έχετε κάνει κάποια ανάλυση σχετικά. Μπορείτε παραδείγματο χάρη να μας ε, πείτε ποια είναι η ε, ανάλυση ελαστικότητας ε, που έχετε κάνει παραδείγματο χάρη πώς θα ε, κινηθεί η κατάσταση εάν είναι τα επιτόκια παραδείγματο χάρη κατά 1% υψηλότερα και για ποιον πληθωρισμό θα μιλούσαμε σε περίπτωση νομισματικής συρρήκνωσης ή λιγότερο ε, ισχυρής επέκτασης. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα, είπατε ότι πιθανώς θα πρέπει να συσταθεί μια bad bank, ε, είπατε κάποια εταιρεία χαρτοφυλακίου, έτσι το κατάλαβα. Το ερώτημά μου είναι ποιος ε, θα αναλάβει τον κίνδυνο είχαμε μία μελέτη του συναδέλφου Χέριχ ο οποίος προειδοποίησε, είπε ότι θα πρέπει αυτά να τα πληρώσει ο φορολογούμενος ε, τους κινδύνους μιας τέτοιας bad bank και είχε ε, μάλιστα προειδοποιήσει περί τυχόν διατάξεων bank πως θα πρέπει να πει, τα επομίζεται αυτά η τράπεζα η οποία έχει την ευθύνη. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, το βλέπετε γιατί δεν είπατε τίποτα για το ποιος θα υπομειστεί τον κίνδυνο. Σας ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση. Η τεχνική υπόθεση για τις προβλέψεις είναι τα βαρχιπρόθεσμα και μασοπρόθεσμα επιτόκια από τις αγορές. Στην αρχή των προβολών αυτών, μάλιστα θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαν να είναι σταθερά τα επιτόκια στη ε, στιγμή που είχαν κατά την προβολή. Και μετά, πριν από τρία χρόνια, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τις προσδοκίες ε, των αγορών. Αυτό δεν μας δεσμεύει για τα επιτόκια. Εμείς είμαστε ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Απλά είπα ότι ε, αν η κατάσταση στην οικονομία και όσον αφορά την ανάπτυξη του πληθωρισμού θα δώσει νέα σημάδια, θα προσαρμοστούμε και εμείς αναλόγως. Έτσι έχουμε κάνει σε όλη την ε, διάρκεια. Αυτό λοιπόν. Δεν γνωρίζω προσωμιώσεις ή αποτελέσματα προσωμιώσεων. Έχουμε κάνει κάποιες προσωμιώσεις σε άλλο πλαίσιο. Το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα των, στις τράπεζες μια αύξησης των επιτοκίων, αλλά όχι στα μακροοικονομικά μοντέλα. Ίσως το έκανε το προσωπικό, δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν γνωρίζω νούμερα σχετικά. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να σας πω πως αυτό το οποίο είπα δεν ήταν υπέρ ε, μιας ε, πανευρωπαϊκής τέτοιας ε, εταιρείας χαρτοφυλακίου η Bad Bank. Στις ομιλίες μου, και έχω κάνει τουλάχιστον δύο προσφάτως, είπα πως ε, αυτό το οποίο είναι κατάλληλότερο θα ήταν ένα ευρωπαϊκό υπόδειγμα εναρμόνισης αλλά μετά οι εταιρείε αυτές ε, να συσταθούν στο εθνικό επίπεδο, αλλά σύμφωνα με ένα ευρωπαϊκό υπόδειγμα, γιατί είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα δεδομένου του μεγέθους ε, των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βεβαίως ε, της υποψίας που έτσι, πέφτει ως σκιά στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Αυτά για να το ξεκαθαρίσουμε. Και όπως ξέρετε, οι εταιρείε ε, τέτοιες ε, χαρτοφυλάκια έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Σλοβενία τουλάχιστον. Και σε άλλες χώρες βεβαίω ε, ανά τον κόσμο. Είναι η συνήθις συμβουλή του Δελτανή Τάφο ότι για να αντιμετωπίσουμε τη μείωση των μη εξυπηρετώμενων δανείων κάνουμε τέτοιες εταιρείε οι οποίες εάν στηθούν σωστά δεν έχουν ε, αρνητικά αποτέλεσμα απλά μας δίνει περισσότερο χρόνο για να δούμε ποια θα είναι τα στοιχεία του ενεργητικού και να προσπαθήσουμε να τα πουλήσουμε και βεβαίως ε, καθώς ε, μετά βελτιώνεται η κατάσταση και έχουμε ανάκαμψη η ανάκαμψη θα αυξήσει τις τιμές των στοιχείων αυτών έτσι ώστε θα προστατεύσει ακριβώς ε, και την εξέλιξη των εταιριών αυτών. Χαρτοφυλακίου, π.χ. στην ε, Ιρλανδία η εταιρεία, εν λόγω εταιρεία, έχει και κέρδη. Οπότε δεν είναι οπωσδήποτε ένα πρόβλημα κατανομής ζημιών. Βεβαίως στις τιμές ε, αρχικής κατανομής υπάρχει μια ζημιά η οποία προφάται από τις τράπεζες όταν δίνουν τα στοιχεία αυτά με μια συγκεκριμένη τιμή. Ναι, ναι, το ερώτημα μου ήταν ποιο θα αναλάβει τον κίνδυνο, λέει ο κύριος Λούκε. Κοιτάξτε εταιρείε αυτές ε, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είναι και δημόσιε ε, και ιδιωτικέ. Ε, στο ΝΑΜΑ, στο ΣΑΡΕΜ, στη Σλοβενία νομίζω είναι τελείως ε, κρατική εταιρεία, αλλά το ΣΑΡΕΠ και το ΝΑΜΑ νομίζω είναι 51% είναι ιδιωτικό το κεφάλαιο και 49% δημόσιο. Αλλά όπω ξέρετε το κεφάλαιο τέτοιων εταιρεών είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τον ισολογισμό που έχουν μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, εκ μέρου των φιλευτέρων, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για το ότι ήρθατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. Έχω δύο ερωτήσεις να κάνω. Η πρώτη είναι η εξής εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη. Αυτό σε γενικές γραμμές και σε ορισμένα κρατημέλη, πόσο μάλλον, πολύ περισσότερο. Και ρωτώ, η ΕΚΤ έχει τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή κάπως το παραγνωρίζει. Η δεύτερη ερώτησή μου ίσως να είναι πιο ενδιαφέρουσα από πλευράς θεωρητικής. Ε, έχει σχέση στην ελεξάρτηση ανάμεσα στις διατροτικές μεταρρυθμίσεις και την παραγωγικότητα. Μπορεί βέβαια κανείς να μετρήσει την παραγωγικότητα με διάφορους τρόπους. Μερικές φορές την μετράμε υπολογίζοντας το λόγο μισθών στην απόδοση. Όμως σε μία μιλία ε, στο London School of Economics ε, και στην Τράπεζα της Ελλάδας υπήρξε μία ομιλία όπου στο τέλος ο μιλητής αναφέρει διάφορα στοιχεία ε, της συνολικής παραγωγικότητας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και όλοι αυτοί οι δείκτες ε, είναι φθήνοντες. Άρα δηλαδή ρωτώ, τι, τι να κάνει η ΕΚΤ για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα της ευθύνουσας παραγωγικότητας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, αν, έχουμε, αν έχουμε κάποια εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, προφανώς και δεν τα έχουμε. Εμείς έχουμε μόνο τη νομισματική πολιτική ως εργαλείο, αλλά δημιουργώντας ευνοϊκή οικονομικές, ε, χρηματοπιστωτικές ε, δυνατότητες. Ε, δημιουργούμε ένα περιβάλλον και συμβάλαμε και εμείς στην ανάκαμψη, η οποία υποτίθεται θα διευκολύνει την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αν δούμε λιγάκι τα στοιχεία του ΟΣΑ, και ο ΟΣΑ, ξέρετε, δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα την αξιολόγηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κάνει αρκετές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ίσως γιατί πιέστηκαν από τις αγορές, από τα προγράμματα, πάντως το έκαναν. Και οι χώρες οι οποίες ε, ε, δεν ήταν ευάλωτες ε, κατά ήταν ευάλωτες κατά τη διάρκεια της κρίσης, αυτές διότι δεν έκαναν ε, τις μεταρρυθμίσεις ε, που έπρεπε να κάνουν και που αναφέρονται στις ε, δημοσίευσεις του ΩΣΑ. Και αυτά δεν διαφέρουν πολύ από τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εγκρίνονται κάθε χρόνο ε, κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αναφέρομαι στις ε, συστάσεις αναχώρα. Η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις πολύ απογοητευτική. Μέσα τόσο εμείς δεν έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία, αλλά το αναφέρουμε συνέχεια ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και μάλιστα στην παρούσα ε, ετήσια έκθεση, στο τετραγωνίδιο 4, σελίδα 41, βλέπουν ότι εκεί γίνεται δική μνήα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα θέλαμε μάλιστα να δούμε εμείς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, υπέβαλε ένα κεφάλαιο σχετικά με τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές πριν από δύο χρόνια και εκεί αναφέρει τον Δούνου του ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστούν όταν υπάρχει ανάπτυξη. Διότι κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις έχουν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις αρνητικές και μόνο αργότερα προκύπτουν τα θετικά αποτελέσματα. Άρα δηλαδή για να εκμεταλλευτεί κανείς την ανάκαμψη θεωρώ ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να ενταθούν οι προσπάθειες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εκ μέρους του ΣΚΟΕ τώρα ο Φάβιο Δεμάζη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο. Αναφερθήκατε στην έλλειψη συνολικού πληθωρισμού, στο χαμηλό επίπεδο του συνολικού πληθωρισμού ε, και το χαμηλό μισθολογικό κόστος. Βλέπετε κάποια σχέση αυτών των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποδυναμώνουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, κρατούν ε, χαμηλά τους μισθούς και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί ως προς τον πληθωρισμό. Από το 2012, 97% των ε, ομολόγων εταιριών ε, από μη χρηματοπιστωτικό κλάδο με βάση κάποια στοιχεία της Euro Intelligence ή κάποιο άλλο φορέα πήγαν σε μερίσματα, σε αγορές ε, και δεν ε, αφιερώθηκαν σε επενδύσεις. Πόσο αισιόδοξο είστε ότι στο πλαίσιο αυτό της τιτλοποίησης ε, θα αφιερωθούν τα έσοδα ώστε να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για να μειώσουμε αυτό το χάσμα παραγωγικότητας. Και σε ό,τι αφορά την έκθεση της διεθνούς διαφάνειας, αναφέρεται στην ε, σύνοψη, η επιτυχία της πολιτικής του ε, Ντράγκη ε, ακολούθησε μετά κάποιες δηλώσεις των Ισπανών και Ιταλών Πρωθυπουργών σε ό,τι αφορά αντίστοιχε μεταρρυθμίσεις, κάτι που δεν ε, μοιάζει τόσο με αυτή τη δηλώση του κ. Ντάιζεμπλουμ για το να μην ε, σπαταλά κανεί τα χρήματα σε γυναίκε ή ποτά. Αλλά σε ό,τι αφορά τι εξελίξει στην Ελλάδα, είχαμε ε, κάποιε συγκεκριμένε ε, πολιτικέ και η, η ΕΚΤΑ έκανε διάκριση μεταξύ τη οικονομική και τη νομισματική πολιτική. Και είπατε ότι εξαιτία ε, της ε, αποφυγής του να δώσετε προνόμια σε μια ε, στο, στον πελάτη στο, στο, ε, λόγω του δικηγορικού απορρίτου είπατε ότι δεν θα ε, υποβάλλετε τη, τα αποτελέσματα αυτής της ε, έκθεσης επικαλούμενη αυτό το δικηγορικό απόρριτο. Ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις. Όπως σας είπα υπάρχουν κάποια είδη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που σε πρώτη φάση έχουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα και μόνο μακροπρόθεσμα αποδίδουν πιο θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι γνωστό και αναφέρεται σε όλες τις σχετικές μελέτες ε, για την πρόοδο και τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι χώρες ε, που υπόκεινταν, ε, σε προγράμματα προσαρμογής ή πιέστηκαν από τις αγορές, αυτό που έκαναν ακριβώς ήταν κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό στην Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα τώρα και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Βέβαια ισχύει ότι οι δικές μας προβλέψεις ε, εξαρτώνται από τέτοιες εξελίξεις μισθολογικού κόστος και άλλων στοιχείων των τοπικών παραγόντων που επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Για να έχουμε μια σταθερή πορεία πληθωρισμού που δεν απαιτεί περισσότερη νομισματική στήριξη, θα πρέπει ο υφέρπον πληθωρισμός, δηλαδή οι τοπικοί παράγοντες ε, του πληθωρισμού και ενισχύουν την ανωδική του πορεία. Και ελπίζουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και έχουμε θετική προοπτική, γιατί μέχρι στιγμής έχει μειωθεί και το χάσμα της παραγωγικότητας. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των μη χρηματοπιστωτικών εταιριών που συνήθως θέλουν ρευστά και χρησιμοποιούν εκδόσεις ομόλογα για να πληρώνουν τα μερίσματα στους μετόχους, όχι τόσο για την αγορά μετοχών. Δεν κάνουν κάτι τέτοιο εμάς όπως γίνεται αλλού, όπου το, το ποσοστό αύξη, ε, αγοράς των δικών τους μετοχών είναι υψηλό. Αυτό όμως δεν συμβαίνει ε, στην Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει περισσότερο σε άλλες χώρες. Πάντως, αν ε, διαχωρίσουμε το συνολικό των ποσοστών σε επιχειρησιακές και σε, σε επενδύσεις ακινήτων, δηλαδή οι επενδύσει μάλιστα στο κατασκευαστικό κλάδο, στο οικοδομικό κλάδο, οι επενδύσει των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί, έχουν αυξηθεί αισθητά το τελευταίο καιρό και μάλιστα έχει φτάσει σε επίπεδα και πριν τη κρίση. Ενώ οι επενδύσει στον οικοδομικό τομέα υστερεί σε σχέση με τα ποσοστά τη αρχή τη κρίση. Οπότε το συνολικό ποσοστό των επενδύσεων δεν έχει φτάσει στο επίπεδο πριν τη κρίση. Άλλες όμως παραγωγικές επενδύσεις εταιριών έχουν ήδη αυξηθεί και μάλιστα αισθητά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να διαχωρίσουμε τα επιμέρους στοιχεία της, των συνολικών επενδύσεων για να δημιουργήσουμε μια πιο ακριβή εικόνα. Πάντως θεωρούμε ότι οι δικές μας πολιτικές και μάλιστα αυτό είναι γεγονό, δεν είναι καν πεποίθηση ότι οι πολιτικέ μα μείωσαν το, το κόστο κεφαλαίου και σε ό,τι αφορά το δανεισμό και το κόστο του μετοχικού κεφαλαίου και δημιούργησαν ένα πιο ευνοϊκό κλίμα για τις επενδυτικές αποφάσεις και ήδη έχουμε ε, ορατά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την τρίτη σας ερώτηση, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι οι αποφάσεις ε, για τις οριστικές νομισματικές συναλλαγές ε, και τη ομιλίες Ντράγκη ακολούθησαν κάποιες επιστολές συγκεκριμένων κυβερνήσεων. Αυτό δεν ισχύει, δεν ε, στείλε καμία κυβέρνηση επιστολή στον πρόεδρο Ντράγκη πριν την αναγγελία της πολιτικής. Ίσως ε, είχατε κατά νου κάτι διαφορετικό, αλλά καμία σχέση με την απόφαση για τις οριστικές νομισματικές συναλλαγές. Όχι, εγώ είπα για μια ε, μελέτη, για μια έκθεση. Ναι, ναι, όχι, γιατί αυτά διαβάσατε από την έκθεση. Από τους πρασίνους, ο Σβέν Welcome, uh, Καλώς ήρθατε κύριε Κωνστάνσιο και καλό Πάσχα εύχομαι. Πρώτα απ' όλα να σας ε, ζητήσω να απαντήσετε στην τελευταία ερώτηση του Φάμπιο Ντεμάζη για το εάν θα δώσετε την εν λόγω μελέτη. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να μοιραστώ τις εξής σκέψεις ε, μαζί σας. Το τέλος του 2015 αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες έγραψαν μια επιστολή στην Κεντρική Τράπεζα για να έχουν διαφορετική μεταχείριση για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις πυλώνα 2 και να ε, μπορέσουν να έχουν κάποια καθοδήγηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολούθησε αυτή την πρακτική μαζί με άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και Επίσης ε, υπήρξε και κάποια μετατροπή σε προτάσεις ε, που υπάρχουν τώρα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έτσι είχαμε μετατροπή δεσμευτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 155 εκατομμυρίων σε κεφαλαιακή κατεύθυνση, τέτοια που είναι λιγότερο δεσμευτικό. Τέτοιες ε, παρεμβάσεις που βασίζονται σε πολιτική και δεν είναι συνήθις εποπτική πρακτική. Ε, γίνουν βεβαίω το ενδιαφέρον ε, διαφόρων ε, ενδιαφερομένων για τις επαφές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό η Διεθνής Διαφάνεια έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δημοσιοποιεί όλες τις συναντήσεις που έχει με ενδιαφερόμενους. Θα κάνετε κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, ε, θα απαντήσετε και στις άλλες συστάσεις ε, της ε, διεθνούς διαφάνειας περί διαφάνειας και λογοδοσίας. Θα με ενδιαφέρει μια απάντηση σημείο να σημείο ακριβώς για την μελέτη που ανέφερε η Περβάνς Μπερές και ο Φάμπιο Ντεμάζη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, για το τελευταίο ερώτημα του κυρίου Ντεμάζη, συγγνώμη το ξέχασα. Πράγματι η απάντησή μας είναι ότι τα έγγραφα αυτά προστατεύονται από το απόρριτο της σχέσης με δικηγόρου με πελάτη και βεβαίω αρθεί αυτό το απόρριτο μπορεί στο μέλλον να έχουμε δυσκολίες για νομικές γνωμοδοτήσεις από άλλες εταιρείες ε, δικηγορικές. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μας ε, και είναι πράγματι επανάληψη των όσων είπατε. Για τις ερωτήσεις του κυρίου Γκίγκολτ. Εμείς δεν κάναμε τίποτα όσον αφορά το ζήτημα αυτό της ε, κατεύθυνσης όπως ίσως ξέρετε, αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας ανακοίνωσης της Κομισιόν ε, σε κάποια στιγμή που έλεγε ότι ακριβώς θα πρέπει να σπάσει ο πυλώνας 2 σε ένα κομμάτι που θα ήταν σκληρός δεύτερος πυλώνας και πυλώνας 2 κατεύθυνση και πράγματι βεβαίως ε, είναι ερμηνεία της ε, Κομισιόν. Δεν είναι δική μας, ε, δεν ήταν δική μας πρωτοβουλία σε αντίθεση με τα όσα είπατε. Ίσως σας είχε ξεφύγει το σχετικό έγγραφο της Κομισιόν, αλλά ήταν σημαντικό έγγραφο για εμάς και ο πρόεδρος Τράγκη αναφέρθηκε σε αυτό το έγγραφο σε μια συνέντευξη τύπου απαντώντας σε μια ερώτηση. Οπότε, ως αποτέλεσμα αυτού του εγγράφου μάλιστα και της ερμηνείας αυτής της Κομισιόν το οποίο ήταν αντιγραφή των όσων έκανε η Τράπεζα της Αγγλίας εκείνη τη στιγμή και δεν είναι τόσο κακή η πρακτική υπό την έννοια ότι έχει σχέση με το NDA, το ελάχιστο ποσό το οποίο διανέμουν σε μερίσματα οι τράπεζες ε, σύμφωνα με κάποια κριτήρια ε, στην οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων ότι όταν δεν έχουν αρκετά κέρδη και υπάρχει κίνδυνος για το επίπεδο κεφαλαίου τότε υπάρχει ε, κάποιος περιορισμός στην διανομή των κερδών και αυτό το οποίο πράγματι επαληθεύτηκε το 2015 ήταν ότι τα επίπεδα αυτά των ποσών NDA ε, που προέκυπταν από την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 4 και τη ΣΥΡΑ οδηγούσαν σε επίπεδα υψηλότερα από ό,τι άλλες ανάλογες διεθνείς τράπεζες. Οπότε υπήρξε η ανακοίνωση της ε, Κομισιόν ε, που ακολουθήθηκε και επιβεβαιώνεται τώρα από τις προτάσεις της Κομισιόν για την αναθεώρηση αυτών των οδηγιών. Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό, για την ε, διεθνή διαφάνεια. Έχουμε απαντήσει σε αυτό έχουν αναφερθεί τα σημεία με τα οποία βεβαίως συμμορφωνόμαστε και εμείς είμαστε υπόλογοι σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο και έχουμε τις πολιτικές μας τις οποίες ε, εγκρίνετε εσείς. Στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας μας έχουμε βελτιώσει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια το επίπεδο διαφανής. Για τις συναντήσεις έχουμε αποκαλύψει όλες τις συναντήσεις των μελών του Δουσού στο, στη σελίδα μας ξεκαθαρά λοιπόν και με διαφάνεια όπως και με την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κυρία Κάπελ. Ε, παρακαλώ οι συνάδελφοι στο δεύτερο γύρο ένα λεπτό ο καθένας. Λοιπόν, η κυρία Κάπελ, τελευταία ομιλητή στον πρώτο γύρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην ετήσια έκθεσή σας ε, του 2016 αναφέρεστε με λεπτομέρειες ε, στο πρόγραμμα δανειοδότησης της ΕΚΤ ε, και ξεκινάτε από τον Απρίλη και αναφέρεστε επίσης και στις θετικέ επιπτώσεις αυτού του προγράμματος. Την προηγούμενη εβδομάδα η ΦΕΔ έκανε μία ανακοίνωση που μας εξέπληξε, δηλαδή ανακοίνωσε ότι ε, θα προβεί σε ξεκαθάρισμα των ισολογισμών, του δικού της ισολογισμού και θέλω να ρωτήσω στην ΕΚΤ προτίθεστε κι εσείς ε, να κάνετε το ίδιο, να μειώσετε το ποσό που προβλέπετε στον προϋπολογισμό σας. Επίσης η ΕΚΤ Δετάρτη ε, ξέφρασε κάποιες προειδοποίησεις για ε, πομφόλιγε στην αγορά κεφαλαίων. Αυτό θα με ενδιέφερε πάρα πολύ η δική σας άποψη. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Βαλέτα, οι Υπουργοί Οικονομικών αναφέρθηκαν ότι ότι και είπαν ότι ε, ένα ευρωπαϊκό εμόλογο δεν τους ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει δική σας η άποψη και με ενδιαφέρει επίσης να μας μιλήσετε και για τη μείωση της αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε τράπεζες ε, και σε κράτη και πώς ακριβώς θα γίνεται η αξιολόγηση κινδύνου των κρατικών ομολόγων. Κάτι άλλο. Ε, είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρει μια ευρωπαϊκή bad bank. Αυτό είναι πολύ θετικό. Το είπε και ο Γερμανός Υπουργό Οικονομικών. Σε εθνικό επίπεδο αυτό, είπατε, είναι ένα καλό εργαλείο εκαθάρισης, η bad bank. Εμένα με ενδιαφέρει να μας ενημερώσετε για την κατάσταση στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει δυσκολίες τον Ιανουάριο ο κύριος Ρέγκλινγκ προειδοποίησε ότι οι αγορές δείχνουν μια νευρικότητα λόγω του υψηλού χρέου και λόγω της κατάστασης κάποιων τραπεζών στην Πορτογαλία. Και ερωτώ εσάς, ε, στην ε, Πορτογαλία σκέφτεστε να προβλέψετε ένα ειδικό εργαλείο, ένα είδος ε, νομισματικού ελέγχου, EMC. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση σχετικά με το μέλλον του μεγέθους ε, των προεπολογισμών, κάτι που έχει προκύψει από το πρόγραμμα των αγορών μας, δεν έχουμε λάβει απόφαση από αυτού. Η ΦΕΔ δεν έχει αναφέρει καμία λεπτομέρεια. Είπε ότι προτίθεται ε, μακροπρόθεσμα σταδιακά να περιορίσει ε, τους προϋπολογισμούς της. Ο δικός μας ο προϋπολογισμός δηλαδή η ορίμανση αυτών που έχουμε προβλέψει ε, θα διαρκέσει κάποια χρόνια που σημαίνει ότι αν αφήσουμε τα ομόλογα και τα άλλα εργαλεία να οριμάσουν και να αποπληρωθούν, τότε αυτό αυτομάτως θα οδηγήσει σε μείωση από τη στιγμή που θα σταματήσουμε τις αγορές κεφαλαίων. Άρα δηλαδή είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να αγοράζουμε ομόλογα μέχρι το Δεκέμβρη και μετά θα δούμε, θα αποφασίσουμε τότε για το μέλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας φυσιολογικός, ε, μια πεπατημένη το να περιορίζεται ο προπολογισμός μειώνεται όταν σταματάνε αγορές ε, ομολόγων και αυτομάτως περιορίζεται ο προπολογισμό. Γιατί ξέρετε, το να πουλήσει κανείς πριν από την ορίμανση των κεφαλαίων και των ομολόγων, αυτό θα οδηγούσε σε μείωση της ε, τιμής ε, των ομολόγων και σε αύξηση όμως της απόδοσης. Και αυτό δεν ε, είναι κάτι που θα το συστήναμε. Πάντως πρέπει να σας πω ότι με τον χρόνο θα υπάρξει αυτή η μείωση του προϋπολογισμού μας. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξουν αυτές οι φούσκες στην Ευρώπη. Και αυτό αφορά την αγορά των ομολόγων, αφορά τις, ε, την αγορά μετοχών, την ε, ε, τον οικοδομικό τομέα. Αυτό ίσως να αφορά κάποιες περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει πιο δυναμική εξέλιξη των ε, τιμών. Όσον αφορά τα ε, ε, εξασφαλισμένα τα ασφαλή ομόλογα, εμείς δεν έχουμε πει τίποτα από αυτό και δεν τα πούμε τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να έχει κατατεθεί από αυτού. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μελέτη της του ESRB, της ε, ε, Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, αλλά ε, δεν αφορά τα ευρωμόλογα, διότι αυτό το ευρωπαϊκό εργαλείο που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων, που αποτελείται από ακαδημαϊκούς, δεν προβλέπει την κοινή ανάληψη κινδύνου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφαλούς ευρωμολόγου. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ δεν έχει κάνει καμία δήλωση από αυτού. Σας ευχαριστώ. Οπότε πάμε στο δεύτερο γύρο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό ο καθένας. Και εσείς παρακαλώ κύριε Αντιπρόεδρε να είστε λακωνικό, ώστε να ολοκληρώσουμε γύρω στις 4.30. Πρώτος ομιλητή από το δεύτερο γύρο είναι ο Γκαμπριέλ Μάτο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον Αντιπρόεδρο Κωνστάσιο. Είναι αμφισβητό ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν και εξακολουθεί να είναι κέριος παράγοντας στην ανάκαμψη, οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε ένα σενάριο σαν το σημερινό, με τη νέα εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και με την καταγερματισμό τη ε, εσωτερική αγορά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Άνωση. Στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΕΚΤ είπε ότι μάλλον θα κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο τα επιτόκια ή ίσω και να ε, μειωθούν ακόμη περαιτέρω. Ποιο είναι ο χρονικό ορίζοντα ε, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το θέμα των επιτοκίων και αν μειωθούν περαιτέρω σε τι χρονικό περιθώριο μιλάμε. Μιλήσαμε για την κακή τράπεζα. Τι γίνεται όμως με τα κόκκινα δάνεια ή με τις ε, καθυστερημένε πληρωμές τη Ιταλίας γιατί είπατε ότι δεν θέλετε μια πανευρωπαϊκή κακή τράπεζα, αλλά αναχώρα. Επίσης, ε, με βάση τις εξελίξεις, ε, τον πληθωρισμό, ε, σε μερικές χώρες έχει ξεπεράσει το 5% και σε άλλες χώρες είναι κάτω του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι μέτρα θα λάβετε προκειμένου να αναχαιτήσετε αυτή τη μεγάλη αστάθεια και τη μεταβλητότητα των ποσοστών και των δικτών. Μάλιστα, με ρωτήσατε για το χρονικό ορίζοντα και πότε αναμένονται αλλαγές στα μέτρα νομισματικής πολιτικής συμπεριλαμβανομένων και των επιτοκίων. Δεν έχουμε αναλάβει δεσμεύσει σχετικά, γιατί έχουμε την ε, ισχύουσα την πολιτική μας που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει κατάλληλη και περιμένουμε οι εξέλιξεις στην οικονομία να ακολουθήσουν το δικό μας βασικό σενάριο και τις προβλέψεις ε, του δικού μας ε, προσωπικού, αλλά δεν έχουμε αναλάβει δεσμεύσει ω προ συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο πλαίσιο. Αν αλλάξουν τα στοιχεία, αν αλλάξουν οι πληροφορίε που θα λάβουμε, αν αλλάξουν τα δεδομένα, φυσικά θα προσαρμόσουμε τον προσανατολισμό τη νομισματική μα πολιτική. Αυτό ισχύει και για το ποσοστό πληθωρισμού 1,5% που συνοδεύτηκε με πιο απογοητευτικό ποσοστό 0,7% για τον βασικό πληθωρισμό, τον υφέρποντο πληθωρισμό. Αλλά ήδη γνωρίζαμε ότι τα επίπεδα του 2% ε, είχαν τεχνικά υποστεί τις συνέπειες ε, ε, της στατιστικής βάσης και των χαμηλών τιμών πετρελαίου. Σε ό,τι αφορά τις εταιρείε χαρτοκεφαλακίου AMC, εταιρείε διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή ε, θα μπορούσαν να παίξουν κατά κάποιο, ρόλο, κατά κάποιο τρόπο το ρόλο της ε, κακής τράπεζας. Αν είχαμε όμως μια ευρωπαϊκή στρατηγική θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε τις συνθήκες αυτές για τις λειτουργίες τέτοιων εταιριών σε όλες τις χώρες. Μάλιστα, ο κύριος ε, Πέτρο Περέιρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω το ρόλο της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και την σύνηση με την οποία αντιστέκεστε στις πιέσεις ε, για να κάμψετε την νομισματική πολιτική. Είναι αξιέπαινη στα στάση Σε Ό,τι αφορά το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της αγοράς περιουσιακών στοιχείων συγκεκριμένων χωρών σε σχέση με χώρες ε, που έχουν ε, πολύ χαμηλότερα ποσοστά, κάτω του μισού. Ε, αυτό όμως, αν παραταθεί, θα αυξήσει τις ανισότητες στην Ευρωζώνη. Φυσικά υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν αυτή τη διαφορά, αλλά σκοπεύετε να λάβετε κάποια μέτρα για να διορθώσετε τη σχετική κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, NPL, ε, πιστεύετε ότι επήγει η λήψη μιας ευρωπαϊκής απόφασης και σε ποιο βαθμό εξαρτάται από μια μεγαλύτερη ευελιξία ή καλύτερη διευκρίνηση ε, των κανόνων και με μια πολιτική που θα εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο αλλά θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και πολύ πιο αξιόπιστη. Σας ευχαριστώ. Για να με καταλάβουν όλοι Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν θα πάω αντίσω στα πορτογαλικά, αλλά στα αγγλικά για να καταλάβουν όλοι. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αγορών περιουσιακών στοιχείων, δεν υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των χωρών. Αυτό που συνέβη είναι ότι έχουμε καθορίσει ένα συνολικό ανώτατο όριο για την έκδοση χρέου, χρεωστικών ομολόγων και μερικέ χώρε όπω η Πορτογαλία που ήδη στο παρελθόν, το 2010-2011, είχαν, αγοράσει ε, είχαν αγοραστεί δικά τους κρατικά ομόλογα έχουν ε, προσθεθεί σε αυτό το συνολικό υπολογισμό και ε, γι' αυτό και έχουν φτάσει στο όριο έκδοσης από έναν εκδότη. Και όσο πλησίαζε το, πλησιάζεται στο όριο, στο υπόλοιπο πρόγραμμα μέχρι το Δεκέμβριο έγιναν αλλαγές ώστε να κρατήσουμε την ισορροπία και να μην ε, υπερβληθεί αυτό το ανώτατο όριο που έχουμε ανά εκδότη. Αυτός ήταν ο λόγος. Και αν ε, εξετάσετε τις ε, χώρες όπως η Πορτογαλία που σε πρόγραμμα προσαρμογής, είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, αν το εξετάσετε συνολικά, με τις υπόλοιπε χώρες. Οπότε δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση με την αγορά περιουσιακών στοιχείων. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα κόκκινα δάνεια, αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα του άτυπο εκοφήν στη Μάλτα και ο αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης στην τελική συνέντευξη τύπου εξήγησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί με την προετοιμασία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε εθνικό επίπεδο. Όχι δηλαδή πανευρωπαϊκή εταιρεία χαρτοφυλακίου διαχείρισης ε, περιουσιακών στοιχείων, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε, πολύ. Επόμενος ομιλητής από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Αναφέρθηκε ήδη μερικές φορές η έκθεση της ε, Διεθνούς Διαφάνειας και η υποχρέωση διαφάνειας της ΕΚΤ. Όμως η έκθεση αυτή ε, δεν συμφωνεί με τις διαφορές ε, λαϊκιστικές δηλώσεις διαφόρων ε, πολιτικών τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε ότι η διοικητής ε, της Κεντρικής Τράπεζας ε, της Ουκρανίας, κυρία κοτερεπα παρετήθηκε μετά από κριτική σειράς ετών η οποία προσπάθησε επί σειρά ετών να κατευθυνθεί μέσω της κρίσης. Έχω λοιπόν τρεις ερωτήσεις για εσάς θεωρείτε πως ε, η κριτική αυτής της κεντρικής τράπεζας αποτελεί μια απειλή για το σύστημα ανεξάρτητων κεντρικών τραπεζών. Δεύτερον, θεωρείτε πως ε, η συμμετοχή της ΕΚΤ ε, στην εποπτεία και στην Τρόικα ε, θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή ε, στο καθεστώς τους ως ανεξάρτητες αρχές και τρίτον τι άποψη έχετε για την Αμερικανική πρόταση νόμου για το ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εξπόστ εποπτεία μέσω ελέγχων παραδείγματος χάρη ή κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Σύντομα. Βεβαίως στον πυρήνα της νομισματικής ένωσης υπάρχει έννοια ότι η κεντρική τράπεζα είναι ανεξάρτητη. Ε, αν δούμε την απόδοση του πληθωρισμού και της οικονομίας στο σύνολό της, ε, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η ΕΚΤ ε, ασκεί μια νομισματική πολιτική η οποία ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις. Και με την επιτυχία που ανέφερα στην αρχική μου δήλωση. Και συνεχίζουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εξομαλύνουμε πλήρως την κατάσταση στην Ευρώπη. Λοιπόν, οι επιθέσεις ε, τώρα κατά των, της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών είναι κάτι το οποίο βεβαίως ε, είναι εναντίον ενός βασικού στοιχείου του ευρωπαϊκού πλαισίου και με ανησυχεί όσον αφορά τώρα τα καθήκοντά μας. Δεν ήταν τυχαίο το ότι στο άρθρο 127 εδάφιο 5 της συνθήκης ε, ήδη από την ε, συνθήκη λοιπόν υπήρχε η δυνατότητα η εποπτεία να ανατεθεί στην κεντρική τράπεζα και δημοσιεύσαμε 2003 ή 2004 αν θυμάμαι καλά ένα κείμενο το οποίο εξέταζε ακριβώς τα υπέρ και τα κατά του να είναι η εποπτεία εντός ή εκτός των κεντρικών τραπεζών. Και το κείμενο ήταν περισσότερο υπέρ. Ε, ένα κείμενο του ΔΣ ε, για το να είναι η εποπτεία στις κεντρικές τράπεζες. Ε, μάλλον υπόψη όλων των παραγωνών. Και πρώτης κρίσης αυτό. Και αυτό το οποίο είδαμε μετά την κρίση ήταν ότι οι χώρες που είχαν την εποπτεία εκτός κεντρικών τραπεζών τελικά επανέφεραν την εποπτεία στις κεντρικές τράπεζες όπως ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ρητά και στον νόμο Dodd Φρανκ είδαμε ότι αυξήθηκαν οι εποπτικές αρμοδιότητες του Fed. Πρόκειται λοιπόν για ιστορικούς και άλλους λόγους ε, που οδήγησαν σε αυτές τις λύσεις όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην Τρόικα δεν ε, είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε ευρωπαϊκή νομοθεσία ή σε κάποια συνθήκη όπως η συνθήκη του ESM. Οπότε συμμορφωνόμαστε με αυτό. Τέλος, δεν ξέρω την εν λόγω αμερικανική νομοθεσία που λέτε, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά αυτά τα οποία διάβασα στις εφημερίδες και σε δύο ομιλίες ε, μελών του ΦΕΔ με κάνουν να ανησυχώ ότι αυτό θα μπορούσε να εισαχθεί ως ιδέα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, Κατλίνα Εβάνα από τους Σοσιαλδημοκράτες. Αν ε, δεν σας πειράζει θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Λοιπόν, όπως ε, διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ε, σταθερή οικονομική ανάπτυξη, αλλά δεν μπορεί παράλληλα να υπάρχει και υψηλή, υψηλό ποσοστό ανεργίας. Διαπιστώνουμε ότι όλα τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδήγησαν στο να υπάρχει μια πολύ εύθραυστη οικονομική ανάπτυξη με βάση τα κριτήρια που ίσχυαν πριν από την κρίση. Η οικονομική ανάπτυξη που μετρήθηκε μετά την εφαρμογή μέτρων ήταν πολύ μετριοπαθής, αυτό τα έλεγα. Ε, μία ερώτηση σχετικά με την εντολή που έχει η ΕΚΤ σε σχέση με την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, την ΦΕΔ. η ΕΚΤ δεν θα έπρεπε να έχει επιπρόσθετες ευθύνες και μια διευρυμένη εντολή που να αφορά και στην ανεργία, στην οικονομική σταθερότητα και στην ανάπτυξη και όχι μόνο στην σταθερότητα των τιμών. Διότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα έπρεπε να υπηρετεί τους πολίτες, να επιτρέπει στους πολίτες και να τους βοηθάει να έχουν πρόσβαση στην ε, δανειοληψία. Νομίζω ότι η διευρυμένη εντολή της ΕΚΤ, αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό στοιχείο της σημερινής συζήτησης. Ε, πάρα πολύ σύντομα θα σας απαντήσω. Πράγματι αυτό υπάρχει στην εντολή και εμείς ε, δεν αμφισβητούμε τη συνθήκη, γιατί η συνθήκη είναι θέμα των κρατών μελών, ε, το κοινοβούλιο, αυτοί αποφασίζουν και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι συμμορφωνόμαστε. Ήταν πολύ μικρή αυτή σύντομη αυτή η ερώτηση εκ μέρους του ΕΛΚ ο κύριος ε, Τόμας Μαν. Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντσιο. Πριν από ένα μήνα είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την ΕΚΤ ε, στην Φραγκφούρτη και εκεί είχαμε μια πολύ επικοδομική συζήτηση. Αλλά έμεινε μια ερώτηση. Έχουμε όλες τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές, μας τις παρουσίασαν. Τώρα η ΦΕΔ λέει εμείς θα μεριμνήσουμε έτσι ώστε να αγοράζουμε λιγότερα κεφάλαια και να αυξήσουμε λιγάκι τα επιτόκια τότε η ΕΚΤΕ θα πρέπει να έχει μια παρεμφερή εξέλιξη. Όχι ακριβώ την ίδια, αλλά περίπου. Ε, και εσεί και κάνετε και κάποιε προσωμιώσει, δηλαδή τι θα γίνει αν. Και αν είχε λάβει διαφορετική απόφαση η ΦΕΤ, τι θα κάναμε εμεί. Πότε θα έρθει η στιγμή όπου θα πούμε ότι πετύχαμε το στόχο μας. Το 2% πληθωρισμός είναι πλέον μέτρο διαρκείας και όχι βραχυπρόθεσμη επιτυχία. Ε, γίνεται λόγος για την κακοφωνία στο ε, Διοικητικό Σύμβουλο της ΕΚΤ. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Όταν όμως προκύπτει μια διαφορετική θέση όπου δεν προκύπτει και μια ε, σαφής πορεία, τότε τίθενται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και πάρα πολύ άλλοι κίνδυνοι. Εγώ δεν λέω να βάλουμε φήμοτρο, κάθε άλλο, αλλά να υπάρχει μια κοινή πορεία για να υπάρχει και εμπιστοσύνη και να μην ε, ενδίδουν οι αγορές. Κατ' ουσίαν αυτό είναι εκείνο που μας ενδιαφέρει, δηλαδή η αξιοπιστία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ερώτησή σας. Ε, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι στην Ευρώπη έχουμε μια ανεξάρτητη νομισματική πολιτική. Εμείς δεν ε, παρακολουθούμε κατά πόδα στη ΦΕΔ και τα επιτόκια της ΦΕΔ. Αν δείτε την περίοδο ύπαρξης της ΕΚΤ υπήρξαν περίοδοι όπου είχαμε τελείως διαφορετικά επιτόκια. Άλλα στις ΗΠΑ, άλλα στην Ευρώπη. Κάθε κεντρική τράπεζα ανταποκρίνεται στις δικές της τις ανάγκες. Ε, η ΦΕΡΠΟΣ, ο ΦΕΡΠΟΝ, πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε και έτσι η ΦΕΔ άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια. Όμως δεν ισχύει αυτό απόλυτα στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου έχουμε διαφορετικά επιτόκια και διαφορετικές πολιτικές. Και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Κάθε χώρα ε, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις ε, προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει εκείνη και με βάση τις εντολές που έχουν οι κεντρικές τράπεζες. Να σας πω επίσης ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει κακοφωνία ε, στις θέσεις, συνολικές θέσεις της ΕΚΤ. Δέστε λιγάκι ε, τις συνδεύξεις τύπου, τις ανακοινώσεις. Εκεί εμείς εκφράζουμε τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στο σύνολό του και επίση μπορείτε και να δείτε και να διαβάσετε τώρα το τι συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβουλίο. Συζητάμε τη νομισματική πολιτική και αν τα διαβάσετε αυτά θα διαπιστώσετε ότι εξ από αυτές τις συζητήσεις προκύπτει μία επικρατούσα άποψη την οποία συμμερίζονται όλοι. Εντάξει, μπορεί να υπάρξουν ε, ε, κάποιες διαφορές, αλλά η πορεία και η γενικότερη θέση είναι απόλυτα σαφής τόσο στις αρχι... στα αρχικά ανακοινωθέντα πριν από συνέντευξη τύπου ή εκ των υστέρων στις εκθέσεις που δημοσιεύουμε. Είναι φυσιολογικό ότι ε, διεξάγονται συζητήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, αλλά σας λέω υπάρχει μια επικρατούσα άποψη που είναι συνεπής και είναι απόλυτα σαφής σε όλα τα επίσημα έγγραφά μας. Σας ευχαριστώ. Και τελευταίος ομιλητής, όχι λιγότερο σημαντικό, βέβαια, ο κύριος ε, Φερνάντε από το από και Δημοκράτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα είμαι λακωνικός, θα περιοριστώ σε μία και μόνο ερώτηση. Στην ασφάλεια καταθέσεων, στην ολοκλήρωση της Τραπεζική Ένωση. Όπω ξέρετε, στο Συμβούλιο οι συζητήσει είναι σε τεχνικό επίπεδο, δεν έχουν φτάσει σε πολιτικό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις για τη σχετική έκθεση. Έχουμε την έκθεση του εισηγητού που ε, προβλέπει μια αλλαγή τη φύση της πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη μετάβαση από ένα μοντέλο πλήρου ε, εγγυήσει, πλήρου ε, ασφάλισης, ευρωπαϊκής των καταθέσεων και το, από το μοντέλο της αντασφάλισης με ελάχιστο επίπεδο αμοιβαίας ανάληψης των κινδύνων ή επιμερισμού των κινδύνων. Αυτή την επιστοδρόμηση στις, ή μάλλον την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις, πώς τη χαρακτηρίζετε, θετική ή αρνητική και θα ληφθεί υπόψη από του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχουμε δημοσιεύσει τη γνωμοδότησή μας επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα εγγύης καταθέσεων, το ΕΝΤΙΣ. Όλα τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτή τη γνωμοδότησή μας και μάλιστα υπάρχει μια καταληκτική προθεσμία το 2024 αν θυμάμαι καλά για την πλήρη εφαρμογή ενός, συστήμα, ενός πλήρου συστήματος εγγύης των καταθέσεων. Και λέμε στο σχολιασμό μας ότι θα θέλαμε όπως συμβαίνει και με το FDIC, ε, να υπάρχει μία γραμμή πίστοσης για συμπλήρωση ε, των πόρων εφόσον χρειαστούν και φυσικά θα τα επιστρέψουμε, όπως συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μιλάμε και για τα χαρακτηριστικά αυτού του ευρωπαϊκού συστήματος. Όλα τα λέμε ξεκάθαρα στη γνωμοδότησή μας και σε αυτήν εμένω. Παρακολουθούμε βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σύστημα αυτό και δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση των συζητήσεων και ποια θα είναι η τελική απόφαση στο Συμβούλιο. Και μάλιστα όταν υπευλήθη η ιδέα της Τραπεζικής Ένωσης ε, είπαμε ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί με έναν μηχανισμό εξυγίανσης και με ένα σύστημα εγγύης καταθέσεων. Αυτή ήταν η θέση μας ε, και ε, εξ αρχής και εμένουμε σε αυτή και τώρα. Αν ε, έχετε ακόμη τρία λεπτά, θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Ντεσάντο στη διαδικασία Catch the Eye για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, αγαπητέ φίλε, είχα πολλέ ερωτήσει, αλλά δυστυχώ χρόνο δεν έχουμε. Γι' αυτό θα περιοριστώ κι εγώ και θα συνεχίσω τον ηρμό του κυρίου Φερνάντε με μία ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύηση Καταθέσεων. Η κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Πορτογαλία ανησυχεί για την καθυστέρηση σε, στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Γιατί είναι πολύ σημαντικός αυτός ο πυλώνας της Εγγύηση καταθέσεων. Ποια είναι τα βασικά εμπόδια, γιατί δεν μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε, επιτέλους να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο τη ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση. Πιστεύετε ότι με την εξασφάλιση και αυτού του πυλώνα θα εγγυηθούμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αν ναι, γιατί δεν επιταχύνονται οι εργασίες ως προς την ολοκλήρωση και αυτού του πυλώνα. Δεν μπορώ εγώ να πιθανολογήσω τις θέσεις ή να εξηγήσω τις αμφιβολίες ή την καθυστέρηση σε ορισμένε χώρες ε, που οδήγησαν σε αυτή την ε, αργοπορία στο Συμβούλιο γιατί υπάρχουν μέτρα μείωσης του κινδύνου και υπάρχουν μέτρα επιμερισμού του κινδύνου. Και εμείς θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν εκ παραλλήλου. Και η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης απαιτεί στη τελική ανάλυση και την ολοκλήρωση και τη συμπερίληψη του συστήματος εγγύης καταθέσεων. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα επιχειρήματα, εμένω στην ανάγκη ε, προσθήκης και αυτού του συστήματος. Θα ήθελα να προσθέσω και ένα άλλο στοιχείο. Το σύστημα εγγύης καταθέσεων είναι σημαντικό ε, και ως εργαλείο ε, δημιουργίας εμπιστοσύνης. Βέβαια δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να αποτρέψουμε κάποιες ε, χρεοκοπίες που θα τραπεζών που θα πετήσουν και πληρωμές. Αυτό δεν συνέβη το και στην κρίση. Αυτό που μας ενδιαφέρει και γι' αυτό χρειάζεται το σύστημα υγιής καταθέσεων είναι να δημιουργήσει εμπιστοσύνη στο νόμισμα και γενικώ στην οικονομία. Και είναι επίση σημαντικό να καταπολεμηθούν κάποιες, να καταπολεμηθούν κάποιες παρεξηγήσεις. Και αυτό θα γίνει με την ε, αύξηση της εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι απαραίτητο και για την Ένωση Αγορών Γιατί ένα από τα εμπόδια σε μια πλήρη Ένωση Αγορών και την αγορά ε, χρεογράφων και κινητών αξιών παντού είναι αυτές οι παρερμηνίες ε, που υπάρχουν για την πιθανότητα μετάδοσης του κινδύνου. Φυσικά πιστεύουμε ότι θα ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η εμπιστοσύνη στις ε, χρηματαγορές στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε και εκ μέρους της Επιτροπής μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας αφιερώσετε δύο ολόκληρες ώρες και μας δώσατε πολύ εύστοχες ε, και έγκριτες παρατηρήσεις για την κατάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά όλους για τη συμμετοχή, για τις εύστοχες ερωτήσεις σας και για την πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση που επίδεξετε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σάιμον για να περάσουμε στο σημείο 5 της σημερινής διάταξης. Okay, dear talks, we go on with point number five, our channel budget of... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε σημείο 5, προεπλογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Ζίγκφριντ Μουρεσάν. Θα κάνει μια γενική εισαγωγή για να ακούσει και τις απόψεις των μελών της Επιτροπής μας. Λοιπόν, πέντε λεπτά ο εισηγητή. μετά ο εισηγητή, ε, ο δικό μα από την ΕΚΟΝ, ε, που επίση πέντε λεπτά λογικά θα μιλήσει. Μετά Νίλ Στόρβαλτ ε, και η Λυπή. Ξεκινάμε λοιπόν με τον εισηγητή τη Επιτροπή Περιπολογισμών. Έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που θα ακούσετε και την άποψη Επιτροπής Προπολογισμών για τον προϋπολογισμό. Να σας πω πως σήμερα ξεκινάω τις επισκέψεις μου στις ε, ειδικευμένε ε, επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου για να παρουσιάσω τις απόψεις μου, τις απόψεις της Επιτροπής μας και βεβαίως για να ακούσω και τις δικές σας προτεραιότητες για τους συγκεκριμένους ε, κλάδους αρμοδιότητός σας. Βεβαίως, πρόκειται για επιστροφή, καθώς είμαι αναπληρωματικό μέλος και αυτής της Επιτροπής ε, και είναι άρα πιο ευχαριστή η σημερινή συνάντηση. Υπέβαλε μια έκθεση για κατευθυντήριες γραμμές για τον προπολογισμό του επομένου έτους ε, που εγκρίθηκε στο Στρασβούργο τον Μάρτιο με ευρία πλειοψηφία και είπα εκεί πως η, η άποψή μου είναι πως οι πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του επόμενου έτους πρέπει να είναι πρώτον ανάπτυξη και δουλειές και δεύτερον η ασφάλεια των πολιτών. Για το πρώτο, ε, ανάπτυξη και δουλειές. Είπα πως αυτή πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα γιατί κατά τα τελευταία δύο έτη όλοι οι πόροι που μπορούσαν να διατεθούν διατέθηκαν για τη μεταναστευτική κρίση. Αλλά βέβαια η οικονομική κατάσταση δεν βελτιώνεται από μόνη τη. Γι' αυτό είπα ότι τώρα είναι η στιγμή να εστιάσουμε περισσότερο στο να ενισχύσουμε την οικονομία μας, να κλείσει το χάσμα των επενδύσεων. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει, ότι θα πρέπει να γίνει, χρησιμοποιώντας αυτά τα οποία έχουμε για επενδύσεις σε καινοτομία, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε νέους επιχειρηματίες, οπότε ήθελα να δω το πρόγραμμα COSME, το οποίο στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον ορίζοντα 2020, την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που ξέρω πως είναι σημαντική και για πολλούς συναδέλφους ε, της Επιτροπής σας. Θα ήθελα αυτά λοιπόν να μπουν στον προπολογισμό του επομένου έτους και βεβαίω συμφωνώ και με την γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ για τα προηγούμενα έτη όπου τονίζεται ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην στήριξη των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για την ασφάλεια, την δεύτερη προτεραιότητά μου, όπως ξέρετε, οι πόροι που έχουμε είναι πολύ περιορισμένοι στον τίτλο 3, γι' αυτό το θέμα είναι πώς θα επιτύχουμε το μέγιστο με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε στην διάθεσή μας. Και οπωσδήποτε τμήμα της απάντησης θα είναι ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών της Ένωσης που έχουν αρμοδιότητα δικαιοσύνης και εσωτερικών, Europol, Eurojust, Frontex, EASO, αλλά βεβαίως και την άμεση γειτονία μας προς Ανατολάς και προς Νότον για του συγκεκριμένου φακέλου τώρα τη ΕΚΟΝ. Ένα, για το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. όπω ξέρετε υπάρχει πρόταση να παραταθεί και να ξεκινήσει το ΕΦΣΙ 2 τον Ιούλιο του 2018. Από τη σκοπιά του υπολογισμού, όπως ξέρετε, η Κομισιόν προτείνει να υπάρξει άλλο 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στην εγγύηση της Ένωσης και να φτάσουμε στα 150 εκατομμύρια από τα αδιάθετα, 500 εκατομμύρια από δημοσιονομικά μέσα και το μέσο συνδέοντας ε, την Ευρώπη και 450 εκατομμύρια από το προσδοκόμενο θετικό ε, αποτέλεσμα. Και βεβαίως προτείνουμε ε, ως Κοινοβούλιο να μην υπάρξουν περικοπές στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη Οπότε οι εισηγητές του Κοινοβουλίου προτείνουν 650 εκατομμύρια ευρώ να χρηματοδοτηθούν από τα αδιάθετα στο ΠΔΠ και 450 εκατομμύρια από το αναμενόμενο συνολικό θετικό αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με, τις, ε, με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα δεσμεύσεων για το FC1, προβλέπουμε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε δεσμεύσεις το 2018 και 135 εκατομμύρια ευρώ στο FC2 το 2018. Τώρα, δεύτερον, για χρηματοδότηση προγραμμάτων όπως το Φισκάλις και Περικλής, χρειαζόμαστε επαρκείς πιστώσεις βεβαίως και για αυτά τα προγράμματα, οπότε και αυτά θα είναι προτεραιότητά μου. Τρίτον, για τις τρεις ε, υπηρεσίες εκείνες οι οποίες εμπίπτουν στη δική σας αρμοδιότητα, Πρέπει να τονίσω ότι οι υπηρεσίες αυτές ε, δεν χρηματοδοτούνται πλήρως από τον προπολογισμό της Ένωσης. Συγχρηματοδοτούνται εν μέρη από τις εθνικές αρχές ε, και εν μέρη μέσω τελών. Οπότε έχουν κάποιες πηγές εσόδων και βεβαίως την επιδότηση της Ένωσης και τα τέλη που χρεώνουν στους χρήστες. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν καλύπτει πλήρως τα έξοδά τους και αυτό είναι σημαντικό όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή η οποία θα πρέπει να μετακομίσει από το Ηνωμένο Βασίλειο σε κάποια άλλη χώρα όταν λάβει χώρα το Brexit και δεδομένου του ότι η Ένωση δεν χρηματοδοτεί την EBA εξ ολοκλήρου Όπω είπα υπάρχει και συγχρηματοδότηση από εθνικέ αρχές και τέλη που χρεώνουν στους χρήστε. Ε, θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη ε, όταν μιλήσουμε για το κόστο τη μετακόμιση. Οπότε δεν θα πρέπει αυτό να πληρωθεί εξ ολοκλήρου από τον προπολογισμό τη Ένωση. Θα πρέπει να δούμε ε, βάσει το τι θα γίνει και με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη μεταβατική περίοδο εάν θα υπάρξει κάποιο κόστος για την μετακόμιση της CBA του χρόνου ή αν θα ξεκινήσουν ε, το τελευταίο έτος μόνο. Τέλος, όσον αφορά τα πιλωτικά έργα, όπως ξέρετε, όλοι οι συνάδελφοι βεβαίως ε, μπορούν να υποβάλουν κάποια πιλωτικά έργα. Εγώ θέλω να υποβάλλετε πολλά για να χρηματοδοτήσουμε τα καλύτερα. Τα σημαντικά μηνύματα είναι τα εξής. Θα μπορέσουμε να περιλάβουμε στο τελικό πακέτο μόνο τα έργα εκείνα τα οποία έχουν προαξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε το μήνυμα προς συναδέλφους είναι ένα. Οτιδήποτε σκοπεύετε να καταθέσετε για προχρηματοδότηση πρέπει να πάει στην Κομισιόν για προαξιολόγηση. Η προθεσμία είναι 3 Μαΐου. Οπότε πρέπει να υποβληθούν για προαξιολόγηση και από τα έργα τα οποία έχουν βαθμολογηθεί καλά από την Κομισιόν, δηλαδή α ή β τουλάχιστον, ε, μετά από συζητήσει με τις πολιτικές ομάδες θα δούμε ποιο θα είναι τα καλύτερα πιλωτικά έργα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι αναμένω την συζήτηση μαζί σας και σήμερα και κατά τη διάρκεια του έτους. Νομίζω είμαστε στην αρχή της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, που δεν υπάρχει κάποιος άλλος παρά μόνο ο μιλητής της Άλντε δεν είναι η πρώτη φορά που προεδρεύω εγώ και είναι η Άλντε η πρώτη η οποία λαμβάνει το λόγο. Ο Νίλ Στόρβαλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται στις διάφορες επιτροπές και υποεπιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει γενική σύμπνοια σε ό,τι αφορά το προϋπολογισμό του 2018. Και όπως είπε και ο κύριος Μαρασάν, οι προτεραιότητες, ε, οι βασικές είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Δεν νομίζω να διαφώνει κανείς. Γι' αυτό είπα ότι οι περισσότερες επιτροπές βρίσκονται στην ίδια ε, γραμμή πλεύσης. Ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστιο επενδυτικό χάσμα. Ξέρουμε ότι οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γεφυρώσει τα χάσματα που υπάρχουν είναι ελάχιστες. Άντε να καλύψουμε μερικά χιλιοστά, αλλά εδώ έχουμε χιλιόμετρα που πρέπει να κλείσουμε, να γεφυρώσουμε. Επίσης, ε, συνεχίζονται οι συζητήσεις για το FC1 και FC2. Το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, στην πρώτη φάση δεν ανταπεξήλθε στις προσδοκίες μας, ό,τι περιμέναμε όταν ξεκίνησε το σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα υψέλθω σε λεπτομέρειες για τις αδυναμίες αυτής της πρώτης φάσης του ΕΦΣΥ. το πρόβλημα ήταν ότι ήταν σχετικά κάποιες ανόητες αποφάσεις ε, και των χωρών και των θεσμικών οργάνων. Ε, και το γεγονό ότι οι αποφάσει για το ΕΦΣΥ πρέπει να είναι ανώνυμες οδήγησε σε μια διαφωνία των κρατών μελών που δεν μπόρεσαν να εγκρίνουν συγκεκριμένα προγράμματα, οπότε ε, είχε μεγαλύτερη ελευθερία στις αποφάσεις και με μεγαλύτερο δικαίωμα. Υπήρχε βέβαια ένα τμήμα σχετικά καλά οργανωμένο, το front loading για, το, για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ήταν ειδικά ιδιαίτερα επιτυχές και υλοποιήθηκε σε σχετικά σύντομη περίοδο. Επίσης, ε, έγινε κάποιες προσπάθειες περικοπής του συνδέοντας την Ευρώπη και συρρήκνωσης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αλλά αν υλοποιηθεί κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει πρόβλημα σε όλους. Δεν το δεχόμαστε γιατί ήδη έχουμε ένα προϋπολογισμό που από διαρθρωτικής πλευράς είναι δορυφορικός ουσιαστικά, με όλο και λιγότερες ελευθερίες και άμα αποχωρήσει και το Ενωμένο Βασίλειο θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι ελευθερίες και οι δορυφόροι θα ξεφύγουν ε, το ελέγχου μας και θα πετάνε αριστερά και δεξιά χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης, ζητούμε επαναφορά των κονδυλίων ε, στον ορίζοντα 2020. Εμείς το λέμε, αλλά δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται. Γιατί το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να περικόψουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάντως, το ορίζοντας 2020 ήταν πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Παρόλο που υπήρχαν κάποιες αδυναμίες και εκεί, στη διάρθρωση, αλλά θέλουμε να αποκατασταθούν τα κονδύλια και να μην συρρυκνωθεί. Πάντως νομίζω όπως είπε και στην αρχή υπάρχει μεγάλη συμφωνία ως προς τον προϋπολογισμό. Τώρα στο Catch the Eye, η συντονίστρια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ε, κυρία Περβάς Περές. Μια και δεν έχουμε άλλους και οδησηγητές, ε, καλό είναι να σεβόμαστε την σειρά των αγοριτών των ομάδων Άμα, σας είχα, άμα είχε ορίσει το κόμμα σας θα το είχα κάνει. Ευχαριστούμε κύριε Μουρασάν που δώσατε έμφαση στα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης και της ε, τόνωσης της απασχόλησης. Συμφωνούμε και ε, στο δεύτερο επενδυτικό σχέδιο γιούνκερ θα έχουν μεγάλη σημασία αυτά τα δύο θέματα και είπατε ότι αρχίζουν και διαφαίνονται κάποιες λύσεις στις συζητήσεις μεταξύ των συνεισηγητών. Και ελπίζω στην έκθεσή σας να συμπεριλάβετε αυτά τα σχόλια και να τα τονίσετε. Εγώ θα σταθώ σε τρία σημεία που είναι πολύ σημαντικά και για τη δική μας Επιτροπή. Καταρχήν, αναφερθήκατε στην ιδιαίτερη κατάσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Όντως, το είχαμε επισημάνει και πέρυσι, ζητώντας ο προϋπολογισμός του οργανισμού αυτού να λάβει υπόψη και το κόστος της μελλοντική απόφασης. Και σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση της ΕΑΤ, η απόφαση αυτή δεν πρέπει να αναβληθεί για το τέλος της ε, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και επίσης θα πρέπει να τηρηθούν και κανόνες ατοδότησης του οργανισμού αυτού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Και καταλαβαίνω ότι θέλετε να τονίσετε τη, τα διάφορα στοιχεία της χρηματοδότησης του οργανισμού αυτού, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως ε, πρόσχημα για να συρρυκνώσουμε τον προϋπολογισμό των οργανισμών γιατί είναι σημαντική οι αρμοδιότητε των οργανισμών και θα πρέπει να έχουν και τα απαραίτητα κονδύλια για να ανταποκριθούν στο έργο τους. Επίσης, δεν θα πρέπει να ανοίξουμε και πάλι το κουτί της Πανδώρας σε ό,τι αφορά την στήριξη που θέλουμε να παράσχουμε στις στις ε, γνωμοδοτήσεις που θα ζητήσουμε για χρηματοπιστωτικά θέματα και από άλλους φορείς. Και θα πρέπει και το έργο τους να γίνεται η... το έργο τους ε, σε, ευνα... σε κατάλληλες περιστάσεις, να μην παρεμποδίζεται, ιδιαίτερα τις Financial Watch και αντίστοιχων φορέων. Και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να βρούμε και αυτή την ισορροπία στην έκθεση. Ευχαριστώ, Περβόνς, ο Άλφρετ. Yes, I, just would like... Ε, θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω τον εισηγητή σε σχέση με αυτό που είπε, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε για τα πιλωτικά προγράμματα, τα πιλωτικά προγράμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά την άποψή σας, ε, είναι δυνατόν να υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης για το Όπω ακριβώς ε, τα πιλωτικά προγράμματα που προέκυψαν από τη βάση του Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πώς εξελίχθηκαν αυτά. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά το τι προτείναμε εμείς. Αλλά μήπως υπάρχει έτσι μια συνοπτική εικόνα για το πώς εξελίχθηκαν αυτά τα πιλωτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια των ετών. Γιατί έτσι θα έχουμε μια καλύτερη ιδέα για το τι μπορούμε να προτείνουμε, να έχει νόημα δηλαδή, και πώς ότι ε, δεν χρειάζεται να προτείνουμε πράγματα τα οποία τελικά αγνοούνται. Ο Σβέν. Πρέπει να πω ότι οποτεδήποτε γίνονται αυτές οι συζητήσεις για τον προεπολογισμό ε, της ΤΙΝΕΚΟΝ υπάρχει δύσπηρασμός, όπως και όταν γίνεται ο προϋπολογισμός ε, στο σύνολο του Κοινοβουλίου. Υπάρχει τώρα το θέμα του, της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και βεβαίω, μπορεί κανείς να αμφισβητήσει κατά πόσον η δομή του προπολογισμού αντικατοπτρίζει τους ε, στόχους του 2020 με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, εξακολουθούμε να δαπανάμε χρήματα για το μίσο που δεν τα πάμε πολύ καλά. Πράγματος χάνει βιωσιμότητα, αντιμετώπιση της φτώχειας, οικονομική ανάπτυξη. Και οποτεδήποτε διαφαίνεται ένα κενό ξαφνικά ε, σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να αναδιατάξουμε τις προτεραιότητές μας. Πρέπει υποτίθεται να γίνει αυτή η συζήτηση, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς τους φορολογούμενους ε, που έχουν δαπανιστεί πολλά χρήματα για μη βιώσιμη γεωργία, πώς είναι δυνατόν να έχουμε χρήματα για να επενδύσουμε σε επενδύσεις με μελλοντικού προσανατολισμούς. Τώρα, όσον αφορά τις δικές μας τις προτεραιότητες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να παραμείνουν αποτελεσματικές. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές πρέπει πράγματι να γίνουν πιο αποτελεσματικές και όσον αφορά ε, την ε, Ένωση Κεφαλαίων και όσον αφορά την, ε, τις προβλέψεις για το μέλλον αφετέρου. Έχουμε συζητήσει με τη Eurostat και με τους νομοθέτες για το μελλοντικό νομοθετικό πρόγραμμα. Το Κοινοβουλίο κατόρθωσε να ορίσει μια ολόκληρη σειρά προτεραιοτήτων και όταν ε, κάνουμε τις καταγραφές του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουμε κατά νου κατά πόσον οι προτεραιότητες ε, για τις οποίες έχουμε ψηφίσει το παρελθόν κατά πόσον αυτές έγιναν δεκτές ε, από τη Eurostat. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι κάναμε πολλή δουλειά για την ε, δημοσιονομική και φορολογική συνεργασία στο πλαίσιο μιας εξεταστικής επιτροπής και διαπιστώσαμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο συνεργασίας ανάμεσα σε ε, νομοθέτες. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι στον προϋπολογισμό για να βοηθήσουμε τους ε, τις αρχές εφαρμογής του νόμου και κυρίως τις ε, αρχές που εργάζονται για τα δημοσιονομικά, νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επένδυση. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν επιθυμεί κάποιος άλλος συνάδελφος ε, να λάβει το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye. Από ό,τι βλέπω όχι. Ως εκ τούτου ε, δίδω και πάλι το λόγο στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, όσον αφορά σχετικά με τον συνάδελφο από την Αλντε, πράγματι πρέπει να βελτιωθεί το εργαλείο ΕΨΗ και νομίζω ότι ε, αυτό ε, πρόκειται και να κάνουμε με το FC2 σε σχέση με το FC1. Τώρα, όσον αφορά τις ε, παρατηρήσεις της κυρίας Περές ε, θα τα καταγράψουμε το 6 δεν θα γίνει του χρόνου, άρα δεν θα, υπάρξει, δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις ε, του χρόνου τουλάχιστον στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χρόνου το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει και δικαιώματα και υποχρώσει. Βεβαίω, εάν οι διαπραγματεύσει για την αποχώρηση τη μεγάλη Βρετανία μα οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές επιπτώσεις στον προπολογισμό όσον αφορά τι διάφορε κατανομές για τι α πούμε, παράδειγμα εταιρείε ή υπηρεσίε που ασχολούνται με τα φάρμακα, τότε θα πρέπει να γίνουν κάποιε προσαρμογέ. Για τα πιλωτικά προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο ε, δημοσιεύει μία έκθεση και εμείς ε, παρακολουθούμε πάντα και την εξέλιξη του πιλωτικού προγράμματος που προτείναμε εμείς. Ε, βέβαια δεν παρακολουθούμε την εξέλιξη πιλωτικών προγραμμάτων άλλων συναδέλφων θεωρώ ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε την Κομισιόν ε, κατά πόσον τελικά αυτή την αξιολόγηση ε, μπορεί να τη στέλνει και σε εμάς ε, και όχι μόνο να τη δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Αν δεν τη στέλνει, να μας τη στέλνει. Αυτή η ετήσια αξιολόγηση τόσο των πιλωτικών προγραμμάτων όσο και των προκατακτικών δράσεων. Υπάρχουν αυτά στο site της ε, Κομισιόν. Προς τον κύριο Γκίγκολτ, Σβέν, είπα ότι οι επενδύσεις στις υποδομές, στην καινοτομία, αυτοί ακριβώς είναι οι τομείς που καθιστούν την οικονομία μας ε, πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, πιο καλά προσανατολισμένη στο μέλλον. Γι' αυτό αυτά πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα του προϋπολογισμού μας. Εάν οι υποδομές είναι καλύτερες, εάν η οικονομία Μα μας βασίζεται περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία, υπάρχει και μεγαλύτερη συνεισφορά ε, προς την ανάπτυξη και προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, μακροπρόθεσμα. Ε, πράγματι, οι πολιτικές που προσανατολίζονται στο μέλλον θα έπρεπε να είναι μια βασική προτεραιότητα του προπολογισμού. Συμφωνώ και επαυξάνω επ' αυτού και επίσης και όλα τα άλλα που αναφέρεται σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, των ΕΖΑΣ. Ε, θα συνεχίσουμε βέβαια τη συζήτηση με την Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια, κατά διάρκεια όλου του έτους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα το χρονοδιάγραμμα για τις ε, περαιτέρω διαδικασίες δεν έχει ακόμα οριστεί. Βεβαίω είναι απόλυτα σαφές ότι στις 24 ε, Μαΐου προβλέπεται από την Κομισιόν να εγκρίνει το σχέδιο του προπολογισμού. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 6. Ε, πρόκειται για τα καλυμμένα ομόλογα. Και εδώ τον λόγο έχει ο κύριος Μπαντ Λούκε. Σήμερα γίνεται, θα γίνει η πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή ΕΚΟΝ σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα ε, νομίζω ότι παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συζήτησε και είπε ότι θα έπρεπε, τον, μάλλον ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015, είπε η Επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα. Και το ίδιο το έκανε και η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Δύο εισηγητές ε, έχουμε και θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο στον κύριο Λούκε για 7 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έχετε λάβει το σχέδιο έκθεσης. Ε, τώρα θα ήθελα συμπληρωματικά προς όσα γράφει η έκθεση και το επεξηγηματικό σημείωμα να πω ποιες είναι οι δικές μου συστάσεις για την δουλειά του Κοινοβουλίου. Πρώτον, οι αγορές για καλυμμένα ομόλογα λειτουργούν καλά με ελάχιστη ευρωπαϊκή ρύθμιση. Ε, ξεπέρασαν πάρα πολύ καλά την οικονομική κρίση, είχαν λιγότερες δυσκολίες από τα κρατικά ομόλογα. Υπάρχουν κάποιες χώρες ε, που θα τις λέγαμε παραδοσιακές αγορές ε, και υπάρχουν αυτά τα μέσα επί αιώνες ε, ήδη αυτά τα μέσα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες σε όλες αυτές τις αγορές το νομοθετικό πλαίσιο έχει αναπτυχθεί σε εθνικό πλαίσιο και είναι βαθύτατα εδρεωμένο και στο εθνικό πτωχευτικό δίκαιο και έτσι προκύπτουν διαφορές στο πλαίσιο των καλυμμένων ομολόγων και υπάρχει και μια κάποια ετερογένεια στο πώς γίνεται ακριβώς η διασφάλιση και έχοντας μιλήσει με διαφόρους επενδυτές εκτιμούν ιδιαίτερα αυτή την ετερογένεια δεν μιλάνε για κατακαιρματισμό της αγοράς, αντιθέτως ε, θεωρούν πως ε, αυτό ακριβώς παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον εντός και εκτός Ένωσης. Οπότε, το πρώτο ερώτημα είναι πρώτα απ' όλα το τι θα ρύθμιζε εδώ πέρα ο Ευρωπαίος ε, νομοθέτης. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια καλυμμένα ομόλογα και ακριβώς επειδή είναι τόσο σίγουρα και τόσο δημοφιλή επενδυτικά μέσα απολαμβάνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση, και θα πρέπει ακριβώς στο νομοθετικό αυτό το πλαίσιο να ευνοηθούν ρυθμιστικά και εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι τα καλυμμένα ομόλογα εξαιρούνται από την ε, BRRD από το μέσο διάσωσης με ίδια μέσα το bail tool από την άλλη θεωρούνται ε, ρευστά στοιχεία ενεργητικού επίπεδου 1 και παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για την στάθμιση κινδύνου. Δεδομένων λοιπόν αυτών των πάρα πολύ θετικών χαρακτηριστικών δεν προξενεί έκπληξη το ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος ακριβής ευρωπαϊκός ορισμός για τα καλυμμένα ομόλογα και η επιτυχία τους έχει οδηγήσει στο ότι έχουν αναπτυχθεί νέες ιδέες για το ότι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με τέτοια καλυμμένα ομόλογα. Ε, τα παραδοσιακά προϊόντα, δηλαδή κάποια μικρά έργα και κρατικά ομόλογα διευρύνονται. Π.χ. προχωράνε τώρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επενδύσεις σε υποδομές. Αυτή είναι μια πρόταση ή ακόμα και καταναλωτική πίστη, δηλαδή κάποια μέσα τα οποία ε, επιτρέπουν κάποιο μεγαλύτερο ρίσκο από ακίνητα και κρατικά ομόλογα και υπάρχει έτσι ο κίνδυνος τα καλυμμένα ομόλογα λόγω της ε, επιτυχίας τους να επεκταθούν και έτσι να νερώσει η έννοια του όρου. Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς να υπάρχει η ανάλογη διασφάλιση, δηλαδή να μην υπάρχουν συστημικοί κινδύνοι αυτά τα προϊόντα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι ο Ευρωπαίος ε, νομοθέτης θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σαφές πλαίσιο ορισμών και στο πλαίσιο αυτό να υπάρχουν κάποια ενιαία κριτήρια τα οποία θα βασίζονται σε κάποιες αρχές ε, έτσι ώστε βεβαίως ε, να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες ε, στο εθνικό πλαίσιο και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί ε, χρεοκοπίας. Λοιπόν, προτείνω να υπάρξει σαφής διαχωρισμός ε, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο των καλυμμένων ομολόγων για να μιλήσουμε ακριβώς για μια νέα κατηγορία επενδυτικών προϊόντων η οποία θα μπορούσε να λέγεται παραδείγματος χάρη European Security Notes και όχι καλυμμένα ομόλογα έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο τα κατέστησε τόσο επιτυχή και να επεκταθεί το πεδίο κάλυψης από την τράπεζα έκδοσης και να μεταφερθεί παραδείγματο χάρη στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή υποδομών αλλά να μην υπάρχει η ίδια ρυθμιστική προτίμηση για αυτά σε σχέση με τα παραδοσιακά καλυμμένα ομόλογα γιατί αυτά τα νέα ομόλογα θα έχουν έναν υψηλότερο βαθμό κινδύνου και άρα δεν θα υπάρχει η δικαιολογία για να υπάρχει η ίδια ευνοϊκή μεταχείριση. Και αναφέρω βεβαίως και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Να πω πως πέρα από την ευρύτερη αυτή ε, κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητο υπάρχει μια άλλη κατηγορία που αφορά χρονική ε, επέκταση είτε μιλάμε για soft bullets είτε για CBTs CPTs, το conditional pass-through, η άμεση επανακχώρηση υπό όρους, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε τόσο έτσι ώστε ο εκδότης να έχει τον έλεγχο ρευστοποίησης γιατί έτσι θα μεταφερόταν ο κίνδυνος ε, από τον αγοραστή στον εκδότη του τίτλου και έτσι θα έχουμε άλλα προβλήματα. Γι' αυτό πρότεινα ένα σχετικά, ένα σχετικά σφιχτό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτος και ο δυσυσυγητής, ο Ζήμφριτ Μωρισάν, που εκπροσωπεί τον Τάριους Ροζάτη. Ευχαριστώ όντως. Ο ο Ντάριος Ροζάτη, ο σκιάδης ηγετής του ΕΛΚ, κολλείεται και μου ανέθεσε να τον αντικαταστήσω και να παρουσιάσω τις απόψεις του. Ευχαριστούμε καταρχήν τον Μπέρν Λούκε για την έκθεσή του. Ο κύριος Ροζάτη είναι γενικώ υπέρ της εκτίμησης και των συμπερασμάτων του Μπέρντ Λούκε ε, για ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα καλυμμένα ομόλογα είναι, είναι η δεύτερη σημασία ε, το δεύτερο σημασία μέσο χρηματοδότησης και χρησιμοποιείται από, πολλά, από πολλούς φορείς. Επίσης στηρίζει την ευρωπαϊκή οικονομία. Είμαστε υπέρ τη προνομιακή του ε, μεταχείριση στον ευρωπαϊκό κανονισμό, γιατί πραγματικά εξασφαλίζονται από υψηλή ποιότητα περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα έδειξαν ανθεκτικότητα στην τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν είναι νέα προϊόντα, δεν έχουν έναν οικουμενικά αποδεκτό ορισμό και ο κανονισμός, ο ορισμός τους αναφέρεται σε πολλούς επιμέρους κανονισμούς και έχουμε ένα πολύμορφο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα σε ό,τι φορά και το επίπεδο ακόμη δημόσιας εποπτείας θα πρέπει να δούμε αν δικαιολογείται να, να ζητήσουμε καλύτερη ολοκλήρωση της εθνικής αγοράς καλυμμένων ομολόγων. Πάντως η ομάδα μας ε, πιστεύει ότι η... καλό θα ήταν να γίνει αυτή η συζήτηση υπ' ευκαιρία της έκθεσης πρωτοβουλίας πριν την υποβολή πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της τυποποίηση και της ευελιξίας. Το ΕΛΚ είναι υπέρ ε, μιας ε, διαφανώ και σταθερής αγοράς καλυμμένων, αξιο... Ε, καλυμμένων ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περαιτέρω τυποποίηση μπορεί να ε, βελτιώσει την ελάχιστη πιστοληπτική ποιότητα αυτών των καλυμμένων ομολόγων και να εξασφαλίσει συνθήκε ίσου ανταγωνισμού. Πάντω, η εναρμόνιση θα πρέπει να στηρίζεται σε υφιστάμενα στήματα και να σέβεται τι εθνικέ αρμοδιότητε. Ένα δυνητικό τέτοιο ευρωπαϊκό πλαίσιο καλυμμένων ομολόγων με βάση τι βέλτιστε πρακτικέ θα πρέπει να είναι γνώμονα για τι διάφορε αγορέ. Αυτή τη στιγμή το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, 90% και υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν και άλλες εθνικές αγορές. Ο κύριος Ροζάτη είναι υπέρ ε, της ε, αρχής που προ... της προσέγγισης με βάση την αρχή που προτείνει ο εισηγητής και έτσι μπορεί να δώσει κάποιους προσανατολισμούς χωρίς ε, να επιβαρύνει τις εθνικές προδιαγραφές. Επίση, είναι σημαντικέ οι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τι προδιαγραφέ τη αγορά και πρωτοβουλίε που θα κατευθύνονται προ την αγορά. Βέβαια, κάποιοι τομεί θα πρέπει να περιγραφούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το θέμα τη υπερβολική εξασφάλιση, για παράδειγμα. Over collateralization. Ο κύριος Ροζάτη θα εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή την κάλυψη και την ε, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των καλυμμένων ομολόγων θα πρέπει να βελτιώσουμε την ασφάλεια δικαίου για τους ε, ε, ασθενέστερους επενδυτές. Και σας ευχαριστούμε, επαναλαμβάνω, για την προσπάθεια και την έκθεσή σας. Ο Άλφρεντ Σάντ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον εισηγητή μας που παρουσίασε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις ε, με τους διοκτήτες. Τα καλυμμένα ομόλογα και ήδη ότι είναι πολύ χρήσιμα, έχουν αποδειχθεί στην πράξη. Είναι μια ευέλικτη μέθοδος για να συγκεντρωθούν ε, κονδύλια και κεφάλαια σε ένα σχετικά διαφανές πλαίσιο. Αυτά μέχρι τώρα έγιναν στο πλαίσιο των εθνικών αγορών. Η Δανία και η Γερμανία θεωρούν ότι είναι καθοριστική σημασία σε επενδυτικά εργαλεία. Έχουμε λοιπόν την πρόταση να ρυθμίσουμε τα καλυμμένα ομόλογα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μια οδηγία και μια νόμιμη αντίδραση θα μπορούσε να είναι η ίδια του Διευθυντή του Γραφείου του Κάρτερ που είχε πει ο Μπερτ ότι έχει σπάσει δεν ξανακολλάει. Η πρόταση λοιπόν τώρα έχει κατατεθεί και πλέον εναπόκειται στην Κομισιόν να συντάξει μια οδηγία να ορίσει ένα πλαίσιο για την Ευρώπη. Πρώτον λοιπόν στην κεφαλαγορά ε, θα ήταν αδύνατο να μην υπάρχει περιθώριο για τα καλυμμένα ομόλογα. Η κεφαλαγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εφαρμόζει μόνο ένα μέτρο που να ταιριάζει όλου. Ε, μπορεί να έχει, να υπάρχουν κάποια κενά. Θα προέκυπταν αυτά τα κενά αν δεν συμπεριλαμβάνονταν και τα καλυμμένα ομόλογα. Δεύτερον, πιστεύω ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι είναι υπέρ μια οδηγία για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα των καλυμμένων ομολόγων. Ε, χρειάζεται λοιπόν να αναγνωριστεί μια εθνική πρακτική που έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Αυτό προκύπτει από τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής και επίσης εκφράζεται και στις συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους που οργανώθηκαν από τον εισηγητή αλλά και από εμένα ξεχωριστά. Τρίτον, αναφέρθηκε ότι αυτή η οδηγία θα ωφελούσε τα κράτη-μέλη που τώρα στην αγορά τους δεν έχουν καλυμμένα ομόλογα παρότι ε, τα ομόλογα, διότι τα ομόλογα είναι υποαναπτυγμένα. Είναι λοιπόν σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Φαίνεται να είμαστε σε σωστό δρόμο, όμως υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί να τους έχουμε κατά νου. Αναφέρθηκαν ε, σήμερα. Ο ένας περιορισμός είναι ότι η οδηγία δεν θα ξαναγκάζει να δίδονται πολλές λεπτομέρειες από τις εθνικές αγορές. Όλοι άμεσα εμπλεκόμενοι μοιάζουν να συμφωνούν ότι θα πρέπει να είναι μια προσέγγιση ε, επί της αρχής, όπως λέει και ο συγκητής, και εγώ συμφωνώ επ' αυτού. Επίσης αναφέρθηκε ότι πρέπει να αποδείτε σημασία όχι στο, στο σήμα covered bond. Ο ορισμός ε, θα πρέπει να είναι σαφής για να είναι και σαφές ότι υπάρχει ε, καλυμμένο ομόλογο. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε είναι στο είδος των κεφαλαίων ε, που θα πρέπει να επιτρέπεται να φέρουν αυτό το σήμα των καλυμμένων κεφαλαίων. Αν θα είναι μόνο ενυπόθηκα δάνεια, ενυπόθηκα και κρατικά ομόλογα ή να περιλαμβάνονται και σκάφη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα θέματα καλύπτονται στο σχέδιο της έκθεσης και στην αιτιολογική έκθεση. Για κάποια τεχνικής φύσεως θέματα είμαι λιγάκι επιφυλακτικός ε, ε, για τους άμεσα εμπλεκόμενους. Δεν είμαι πεπισμένος ότι στο σχέδιο ε, είναι σωστή αυτή η πρόταση να υπάρχει παράλληλα και με τα καλυμμένα ομόλογα μια άλλη πρόταση για ευρωπαϊκά ομόλογα εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός χρόνος ορίμανσης. Σε γενικές γραμμές ε, θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή βάση για να υπάρξουν ε, περαιτέρω συζητήσεις. Και πάλι συγχαίρω τον εισηγητή γιατί την πολύ καλή δουλειά και προσβλέπω στην ολοκλήρωση της έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Ευχαριστούμε τον Αλφρέντερ. Καταρχά, θα έπρεπε να έχουμε τώρα την εκπρόσωπο των φιλελευθέρων, αλλά δεν είναι εδώ, γι' αυτό θα λάβει το λόγο ο κ. Μιγκουέλ Βιέγκας, εκ μέρου της ε, Γκουα, που κι αυτός όμως δεν είναι εδώ και δεν εκπροσωπείται, ο κύριος Σβέν Κίκλουτ για τους Παρασύνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί ήταν πολύ συνεργάσιμος στην συνεργασία του με τους και οδησηγητές ε, κατά την εκπόνηση της έκθεσής του. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Γενικώ ε, ακολουθούμε την ίδια γραμμή πλεύσης. Θεωρούμε ότι υπάρχουν σίγουρα πολύ σοβαρότερα προβλήματα στους ευρωπαϊκούς ε, χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς και στις κεφαλαίου αγορές Ευρώπη από την ρύθμιση των ε, καλυμμένων ομολόγων. Δεν υπάρχουν ε, ισχυρά τεκμήρια αυτή τη στιγμή, ούτε για σοβαρότερου κινδύνου για του επενδυτέ ε, η αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη η διευθέτηση αυτού του ζητήματος τώρα. Εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια τη Ένωσης Κεφαλαγορών έχει νόημα να επιφέρουμε κάποιε διευκρινήσει να αποσαφηνίσουμε το θέμα και να βοηθήσουμε αυτό το επιτυχές μοντέλο και πρότυπο να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα στο μέλλον. Πάντως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό το θέμα του σήματος. Ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην αφήσουμε πολλά είδη περιουσιακών στοιχείων να καλύπτονται από τα καλυμμένα ομόλογα, γιατί στο μέλλον ε, έχουμε κάποιου ε, κάποιους που δεν διαπιστώσαμε μέχρι στιγμή. Γι' αυτό προτιμώ μια πιο επιφυλακτική και συνετή προσέγγιση. Πάντως ε, αυτό είναι δεδομένο και ήδη υπάρχουν σημάδια ότι μπορούμε να έχουμε προσεκτική, προσεκτική προσέγγιση και ξεκάθαρο ορισμό. Τότε θα έχει νόημα και μεγαλύτερος εξευρωπαϊσμός η μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτού του θέματος. Πάντως, στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να ζητήσουμε γιατί τα καλυμμένα ομόλογα ε, υπολογίζονται στο πλαίσιο των ε, συνεισφορών προ τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εξυγίαση και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίαση, αφού δεν χρεοκοπούν ποτέ, αφού δεν αθετούν ποτέ τι υποχρεώσει Γιατί περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού, γιατί αν θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτά τα μέσα, θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε από τη βάση υπολογισμού. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και μάλιστα πολύ σοβαρά. Θα ήταν ένα επιπλέον έναυσμα για ένα μοντέλο χρηματοδοτικό που έχει λειτουργήσει πολύ καλά μέχρι τώρα και επίσης θα είναι και μια χρήσιμη συζήτηση για το ποια είναι η βάση υπολογισμού για τη συμβολή, για τη συνεισφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίασης. Και μάλιστα για το θέμα αυτό έχω πολλά και διάφορα να πω. Πάντως θεωρώ ότι είναι πολύ επικοδομητικός ο τρόπος συνεργασίας και υπάρχουν και πολλά κοινά σημεία και πολλά σημεία σύγκλησης. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα ύφους. Μήπως θα έπρεπε ε, να ξεκινήσουμε με το δύο, με το προειδοποιεί, γιατί αν έχουμε από την αρχή τέτοιες προειδοποίησεις, ίσως είναι υπερβολικό δεν είναι θέμα ουσίας, είναι περισσότερο θέμα ύφους και συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των μελλοντικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επαναλαμβάνω, είναι θέμα τυπικό, περισσότερο θέμα ύφους. Ελπίζω να συνεχίσουμε την καρποφόρα μας συνεργασία στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Φωνστόρχ για το EFTD δεν είναι εδώ. Οπότε έχουμε Χάνεμανς για το ENF. Θα μιλήσω Ολλανδικά λοιπόν. Εγώ και το ΙΕΝΕΦ θα δούμε την έκθεση βεβαίως χωρίς ε, κάποια προκατάληψη παρά τα όσα είπε ο κύριος ε, Κίγκολτς γιατί δεν είμαστε υπέρ μιας ε, εναρμόνισης και αντικατάστασης του εθνικού από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Παρόλα αυτά θεωρούμε πως οι διασυνοριακές επενδύσεις σήμερα δουλεύουν μια χαρά μέσω του εθνικού πλαισίου. Γι' αυτό περιοριζόμαστε νομίζω καλύτερα σε μια εθνική, σε ευρωπαϊκό ορισμό και την διαφάνεια των αγορών αν βεβαίως παραμείνει η έκθεση ως έχει και δεν ε, καταλήξει τελείως διαφορετική με πράγματα τα οποία ακούσαμε σήμερα, τυποποίηση, level playing field και ακόμα και ολοκλήρωση ακούσαμε στην Τράπεζα Κεφαλαίου Αγορών. Αν όλα αυτά λοιπόν δεν αλλάξουν τελείως ε, το ύφος και το περιεχόμενο της έκθεσης, τότε μάλλον πιθανότατα θα την ε, εγκρίνουμε. Και θα έπρεπε, κατά αναλογία προς αυτή την έκθεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς να περιορίζεται σε διαφάνεια και στα απολύτως ελάχιστα. Και θα ήταν νομίζω και πολύ χρησιμότερη η Ένωση έτσι. Σας ευχαριστώ κύριε Άνεμαν στην διαδικασία ΚΕΤΣΙΑΙ. Έχουμε την κυρία Περβάνος Μπερές. Ευχαριστώ. Έχουμε εδώ μία πολύ συγκεκριμένη δομή. Και το είπε και ο εισηγητής, πρόκειται για προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται με το ίδιο τρόπο στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχει μια ανισότητα προς τη χρήση τους. Οπότε το θέμα είναι θα, κάνουμε, θα δημιουργήσουμε ένα εργαλείο, ένα μέσο που θα το χρησιμοποιούν παντού. Άρα θα αφισβητήσουμε το σύστημα ή θα ευνοήσουμε τη συνύπαρξη μεταξύ των καλυμμένων ομολόγων και άλλων μέσων. Από ό,τι κατάλαβα, η ιδέα του εισηγητού είναι μάλλον προς τις συνύπαρξεις, αλλά τότε θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Μήπως έτσι μέσω της έκθεσης αυτής ε, τασόμαστε υπέρ του α ή β παραγόγου ή μέσου. Φοβάμαι ότι αν δεν επέμβουμε στην αγορά των καλυμμένων ομολόγων, θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ένα καλό επίπεδο διαχείρισης κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είμαι σίγουρη ότι... Δεν είμαι σίγουρη ποιε θα είναι οι προτάσει ε, του Σουέν Γκίγκολτ. σω θα έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αλλά αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με την ε, ομάδα διαπραγμάτευση, δηλαδή για το κατά πόσο θα πρέπει να ενισχύσουμε ή όχι τι λειτουργίε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας για τα προϊόντα αυτά και αν ναι, υπό, ποιε, προποθέσει. Ευχαριστώ, Περφάνς κάποιος άλλος ε, συνάδελφος θέλει τον λόγο. Όχι. Οπότε τον λόγο έχει ξανά ο εισηγητής. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοδομητική και θετική αντιμετώπιση της έκθεσης. Νομίζω ότι δεν έχουμε μεγάλες διαφορές απόψεων. Γι' αυτό θα είμαι και σύντομος όσον αφορά τις στάσεις της ε, EBA κλείνω περισσότερο να ε, επανέλθουμε στις αρχές ε, οι οποίες διέπουν τα καλυμμένα ομόλογα, δηλαδή να είμαστε πολύ προσεκτικοί και μετρημένοι στην έκθεση σε μια μελλοντική οδηγία και να λάβουμε μέτρα τα οποία θα πηγαίνουν προς μια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ πως ε, τα πράγματα αυτά ουσιαστικά ανήκουν ε, στο εθνικό πεδίο. Το ίδιο και για την εποπτεία. Για να απαντήσω στην ε, Περβάνς Μπερές. Αν δηλαδή το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι εθνικό και έχει στενή σχέση με την εθνική νομοθεσία περί ε, φερεγγαιότητας και χρεοκοπίας θα πρέπει να έχει κάποιο προβάδισμα. Όσον αφορά τα European Secured Notes και τις ε, παρατηρήσεις του Alfred Sand, ε, τις αντιλαμβάνομαι. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι το προϊόν έτσι μπορεί από μόνο του να πετάξει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε μια τέτοια κατηγορία προϊόντων και νομίζω θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης έκθεσης ή νομοθετικής ε, διαδικασίας. Εγώ θα ήθελα ακριβώς να τονίσω την διάκριση μεταξύ των παραδοσιακών καλυμμένων ομολόγων που θα πρέπει να διατηρήσουν αυτόν τον τίτλο και λοιπόν δυνατοτήτων ε, από τις οποίες μπορούμε να διδαχτούμε του πώς θα μεταφέρουμε αυτές τις αρχές σε άλλους τομείς, χωρίς να σημαίνει ότι τώρα θέλουμε τέτοια νομοθεσία. Απλά προδιαγράφουμε, θα έλεγα, το μέλλον και έχει το δικαίωμα ο συνομοθέτης να τα δει αυτά στο μέλλον. Η παρατήρηση του Σβεν Γκίγκολτ με βρίσκει σύμφωνο το ότι θα πρέπει δηλαδή να δούμε την βάση υπολογισμού. Πράγματι τώρα δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι κάτι το νομοθετικό. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Πώς δηλαδή θα υπάρξει αυτή η βάση υπολογισμού, από τι θα αποτελείται, αν θα πάρουμε ή θα καλύψουμε ή όχι τα cover bonds. εδώ πέρα φτάνουμε στα όρια της έκθεσης ε, ιδίας ε, πρωτοβουλίας και ίσως θα πρέπει να πάμε παραπέρα. Λοιπόν, για την ε, αμοιβεοποίηση και αυτό το οποίο είπε ο Ζίγκφριντ Μόρεσαν, την υπερβολική αυτή ε, ναι, εξασφάλιση ε, δεν, δεν ήθελα τώρα εγώ σε αυτή την έκθεση να επεκταθώ περισσότερο για αυτή την υπερβολική διασφάλιση και την αξιολόγηση των αντικειμένων αυτών. Δεν θέλω ούτε να πω πώς θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Εξακολουθώ να θεωρώ την υπόθεση του εθνικού νομοθέτη. Βεβαίω πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εθνικές ε, αγορές ακινήτων. Γι' αυτό θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωπαίος νομοθέτης πρέπει να μείνουμε μακριά. Γι' αυτό ακριβώ εδώ πέρα το ερώτημα του ΕΛΚ για περισσότερες λεπτομέρειες για την υπερβολική διασφάλιση ε, έρχεται σε αντίφαση με αυτό το οποίο είπε και το ΕΛΚ ότι ε, πρέπει αυτά να μείνουν στο εθνικό επίπεδο και να διατηρηθεί ευελιξία. Οπότε συνολικά δεν βλέπω μεγάλες ε, διαφορές ε, και χαίρομαι για τη συνεργασία που έχουμε με τους ε, συναδέλφους και για την ευκαιρία που έχω να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάσταση απολογιών είναι 27 Τετάρτου. Θα τη συζητήσουμε στις 29 Πέμπτου. Στις 3 ε, Ιουλίου θα γίνει η ψηφορία στην Ολομέλεια. Στα διάφορα δεν υπάρχει τίποτα που σημαίνει να σας επισημάνω ότι την επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 24 Απριλίου. 3 με 6.30. Λύει τη συνεδρίαση.